Chers collègues, si vous voulez bien prendre euh, place, que nous puissions... Euh, Καθίστε σας παρακαλώ για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Στο σημείο 20 η ησυχία. Θα δώσω την, το λόγο στον ε, Τόμας ε, Μαν ε, για τις υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια της Ένωσης και την κατάργηση της οδηγίας 96-67. Ο εισηγητής μας παρουσιάζει τη γνωμοδότησή του. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη και αναφέρεται εις ε, τις ε, διάφορες υπηρεσίες ε, τόσο για τα εμπορεύματα όσο και για τους επιβάτες ε, ε, υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να είναι ποιοτικέ και η ποιότητα των υπηρεσιών δεν μειώθηκε διότι δεν υπάρχουν τα σωστά άτομα αλλά διότι από το 96 έχει ξεκινήσει μία φιλελευθεροποίηση οπότε είχαμε καταρτήσει μία γνωμοδότηση όπου λέγεται ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός και θα, να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός κανείς από εμά δεν θέλει μονοπόλια αλλά όταν υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει και ε, μία δίκαιη αντιμετώπιση και να μην το παρακάνουμε. Γι' αυτό και ε, ε, έχουμε απευθυνθεί στην πρόοδο και δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι ηγούνται της ε, του θέματος αλλά κάνουμε μία γνωμοδότηση ε, και ε, έχουμε αναφερθεί εις την εγγύηση των θέσεων εργασίας ένα βασικό άρθρο είναι η αξιολόγηση της κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών και με την Επιτροπή Μεταφορών έχουμε αναφερθεί στην στην εγγύηση των θέσεων εργασίας και στην ε, ε, μετεκπαίδευση. Και είδαμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη οι μισθοί έχουν μειωθεί και ότι τώρα υπάρχει μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φιλελευθεροποίηση λέγοντας ότι χρειάζεται και περαιστέρω απελευθέρωση να υπάρχει και ένας τρίτος επιχειρηματίας που να προσφέρει υπηρεσίες εις ε, το, τα αεροδρόμια με πάνω από 5 εκατομμύρια και 100.000 ε, τόνους που να διακινούνται από το αεροδρόμιο αυτό γι' αυτό και ε, επειδή ε, είχα διάφορες εμπειρίες από αεροδρόμια όχι μόνο στην ε, Γερμανία αλλά και στο εξωτερικό είδα ότι η τιμή της διεκπαιρέωσης αυξήθηκε, οι μισθοί μειώθηκαν και αυτό οδήγησε ότι σε πολλά κράτη-μέλη αυξήθηκαν οι ώρες καθημερινής εργασίας, τα διαλύματα μειώθηκαν και σε πολλά αεροδρόμια υπάρχουν ε, ε, βάρδιες ε, οι οποίες δεν αμείβονται πλέον για επιβεβαρημένη εργασία και υπάρχουν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους εργαζομένους. Πώς θέλουμε λοιπόν και γιατί θέλουμε να υπάρχει βελτιωμένη ποιότητα για να υπάρχει ασφάλεια περισσότερο και για μας σαν ε, πιβάτες αλλά και γενικότερα διότι διαφορετικά θα λέγαμε αν έρθουν με περισσότεροι που θα προσφέρουν υπηρεσίες ε, τότε θα είναι χαμηλότερες οι τιμές αλλά πρέπει να γνωρίζουν και τις διαδικασίες χρειαζόμαστε άτομα τα οποία ταυτίζονται με τη θέση της εργασίας τους και ξέρουν ε, τι χειρίζονται δηλαδή χρειαζόμαστε ένα άλλο θέμα είναι η διακίνηση και το προσωπικό εδάφους, διότι το θέμα είναι τι γίνεται, υπάρχουν καθυστερήσεις και έχω στείλει μία γραπτή ερώτηση ε, εάν όντως οφείλεται η εξυπηρέτηση εδάφου στα αεροδρόμια για την, ε, τις καθυστερήσεις και ο Επίτροπος Κάλλας είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη-μέλη που να εξηγούν και να δικαιολογούν ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στο προσωπικό εδάφους και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση και αργότερα υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Μήπως θα πρέπει να έχουμε έναν κανονισμό γιατί ξέρουμε ότι ε, ε, ε, υπάρχει σε, στην περίπτωση κανονισμού ακριβής εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Γιατί δεν επαρκεί δηλαδή η οδηγία. Γιατί γενικώ παντού χρειάζεται εγγύησης και αυτό θα μπορούσε να προβλεφθεί αλλά πουθενά δεν λέγεται ότι προδιαγράφεται ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση και θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα περισσότερες υπηρεσίες οι οποίες να μας εγγυούνται την ασφάλειά μας. Επίσης είχαμε οργανώσει στην Επιτροπή Απασχόλησης μία ακρόαση με διάφορες ε, αεροπορικές εταιρείες ε, και με εκπρόσωπο του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων και τα απορίσματα της ακροάσεως αυτής προσπάθησα να τα εσωματώσω στην έκθεσή μου και προσβλέπω στη συζήτηση την οποία θα κάνουμε εδώ και θα ήθελα όχι μόνο με τους ε, σκιώδεις αλλά με όλους να συνεργαστούμε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρξει μια κοινή έκθεση την οποία όλοι να μπορέσουμε να στηρίξουμε στηρίξουμε. Ευχαριστώ η κυρία Στένρουκ και μετά ο κύριος Βάκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τόμας Μαν. Πρέπει να σου πω ότι όντως η έκθεσή σου είναι εξαιρετική και οι θέσεις τις οποίες παρουσιάσεις είναι τέτοιες ώστε μπορώ να σε ακολουθήσω σε γενικές γραμμές και είμαι πολύ ευτυχής που η πρόεδρος της Επιτροπής και τα άλλα μέλη επενέβησαν για να μπορεί να παρέμβει στο θέμα αυτό η Επιτροπή Απασχόλησης που είναι πολύ σημαντική για τους εργαζομένους. Τα θέματα τα οποία υπάρχουν εδώ είναι σημαντικά. Είδαμε τις τελευταίες ε, ε, απελευθερώσεις παντού όπου υπάρχει ε, πίεση ανταγωνιστική η οποία επιβαρύνει τους εργαζομένους οδηγεί σε μειώσεις μισθών μέχρι 25% σε όλα τα κράτη-μέλη και εδώ δεν μιλάμε για ένα μόνο ο κράτος αλλά για τα αεροδρόμια ολόκληρη ολόκληρης της Ευρώπης και για θέματα τα οποία προέκυψαν στο παρελθόν. Βάσει λοιπόν της εκπαιδεύσεως, της εκπαιδεύσεως μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και στην ασφάλεια αλλά και γενικότερα. Χρειαζόμαστε σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό εδάφους το οποίο θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των, ε, της ε, εναερίου κυκλοφορίας και και θα μπορέσει να ε, κατανείμει καλύτερα τα βάρη. Αυτό που θέλω να προσθέσω πολύ γρήγορα είναι ότι σίγουρα θα χρειαστεί να συζητούσουμε για το ποιες υπηρεσίες πρέπει να μας εξασφαλίσουν ε, εχέγγυα τα τρόπον ώστε να μην μοιραστούν οι εργαζόμενοι σε δύο τάξεις εργαζομένους πρώτης τάξεως και δευτέρας τάξεως υποδέστερης. Θα πρέπει να να εξασφαλίσουμε να υπάρχουν σωστές συνθήκες εργασίας με σωστή κοινωνική πρόνοια και αμοιβή διότι διαφορετικά ο, βεβαίως στην εναέρια κυκλοφορία το πρώτο μέλημα δεν είναι ο ανταγωνισμός και η μισθή πρέπει να έχει ενισχυθεί η παιδεία θα πρέπει η μετεκπαίδευση να βασιστεί σε γενικώς δεσμευτικές προδιαγραφές ε, διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Τώρα κανονισμός ή οδηγίας. Ε, συμφωνώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε διότι η οδηγία ε, δεδομένη της κατάστασης και της, διαφορετικάς, της διαφοράς στοιχείων θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου να είναι πιο χρήσιμη και γι' αυτό θα ήθελα να καταλήξουμε σε μία κοινή θέση, να μην υπάρχει πίεση ανταγωνιστική ε, προς τους εργαζομένους και να υπάρχουν υπηρεσίες καλού επίπεδου. Ο κύριος Μπάκα και μετά ο κύριος Έντελ. Ευχαριστώ Τόμας. Ε, ε, μπορώ απλώς να συμφωνήσω με αυτά που είπε η Γιούτα Στάινμπρουκ. Έχεις καταρτήσει μια πολύ καλή έκθεση και ε, οι ευχές οι οποίες εκφράστησαν καλύπτουν και το άρθρο 50. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ότι έχουμε σωστά παρέμβει τώρα όσον αφορά την απελευθέρωση ξέρετε ποια είναι η θέση μου δεν είμαι κατά του ανταγωνισμού που προωθεί την καινοτομία και περισσότερη ποικιλία προσφοράς αλλά πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός ισχύει και αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες εδάφους δεν είναι πια μονοπόλια τα οποία δεν ανοίγουν και δεν κινούνται επιτρέπεται ο ανταγωνισμός και πρέπει να προωθηθεί αυτό ούτως ή άλλως αναφέρθηκε και στην Επιτροπή Μεταφορών γι' αυτό και η Επιτροπή μας προσπαθεί να προχωρήσει πέραν των προτάσεων της Επιτροπής Μεταφορών και ε, μας είπε επίσης που νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν εξοικονομήσεις. Σχετικά με τα άρθρα, νομίζω ότι το θέμα του προσωπικού είναι πολύ σωστό έτσι όπως το περιγράφει σχετικά με την παιδεία και την μετεκπαίδευση διότι νομίζω ότι πρέπει για την κατάρτιση να βασιστούμε βάση, ε, στις ε, ανώτατες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και όχι στις ελάχιστες. Αυτό ισχύει και για τους συνεργάτες στα αεροδρόμια αλλά και για τους ε, επιβάτες. Θα πρέπει νομίζω να επιμείνουμε ότι δύο μέρες καταρτήσεως δεν επαρκεί και θα πρέπει να το αφήσουμε στη διάκριση των κρατών μελών διότι κάθε αεροδρόμιο έχει τα, ε, τις ιδιομορφίες του και γι' αυτό πιστεύω ότι όπως ε, και η κοινωνική πρόληψη θα πρέπει να είναι της αρμοδιότητας των κρατών μελών διότι εξαρτάται από τα κυρίαρχα κράτη. Ε, πιστεύω λοιπόν το αν θα είναι οδηγία ή κανονισμός εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι οδηγία για να υπάρξει βάση της αρχής επικουρικότητας μεγαλύτερη επέμβαση των κρατών μελών. Κατά τα άλλα σε συμφωνώ, σε, σε συγχαίρω και σε στηρίζω και πιστεύω ότι θα πρέπει στο μέλλον να υπάρξει και μεγαλύτερη απελευθέρωση στον τομέα των αεροδρομίων ο Τόμας Χάντελ και μετά ο κύριος Μπέκερ. Ε, όταν ένας ε, εκπρόσωπος της Ηνωμένη Αριστεράς ομολογεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, ε, ε, το, διάβασε χαλαρά την έκθεση του, ενός εκπροσώπου του ΕΛΚ δεν θα με πιστέψει κανείς και όμως έτσι είναι διότι αυτό το οποίο παρουσίασε ο Τόμας Μαν βάσει της μακράς προεργασίας και πέραν των κομματικών περιορισμών με βρίσκει σύμφωνο και θέλω όμως να κάνω μία-δύο παρατηρήσεις που αναφέρονται στη συζήτηση που είχαμε μέχρι τούδε διότι ήδη ενισχυμένα και γι' αυτό απευθύνω μία παράκληση στην Πρόεδρο να επιμείνει και στις άλλες επιτροπές θα πρέπει εμείς όπως είπα να επιμείνουμε και να απαιτήσουμε να έχουμε ε, ενισχυμένη εμπλοκή στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων διότι μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών και της δικιά μας το, μας αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και των μισθών. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτούμε κατά πόσο μπορούμε να σκεφτούμε να επέμβουμε και πάλι κατά τρόπον ώστε η αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά να επανέλθει ή στην Επιτροπή μας. Αυτό και τίποτα άλλο. Ένα άλλο σχόλιο και μία πρόταση σχετικά με την τροπολογία 17 αυτής της ε, ε, εκθέσεως. Θα παρακαλούσα να την ξανασκεφτούμε διότι η επιδίνωση των συνθήκων εργασίας και ε, ε, των μισθών οφείλεται σε μια αλλαγή ε, καταστάσεως. Δηλαδή εάν η εργαζόμενοι περάσουν από μια ε, ε, επιχείρηση σε μια άλλη και ίσως εδώ θα έπρεπε να επιμείνουμε ε, να υπάρχει μια ρύθμιση σταθερή η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει το πνεύμα του άρθρου 13α κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μια παρεμφερής ρύθμιση και εδώ για την μεταφορά του προσωπικού από μία επιχείρηση σε μία άλλη. Αυτά είχα να σας πω και τελειώνω. Πριν δώσω το ρόγο στον κύριο Μπέκερ, θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι μιλάμε για το ίδιο θέμα διότι είπατε ότι δεν σας άρεσε η κατανομή των θέσεων με την Επιτροπή Μεταφορών ενώ είμαστε συνδεδεμένη Επιτροπή, είμαστε δηλαδή ε, ε, απόλυτα συνδεδεμένη και σχετικά με το εκτιμώντας 31 και μία ολόκληρη σειρά άρθρων μέχρι το 40 ε, παρεμβαίνουμε πλήρως. Θεωρείται ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι αρκετά πλήρης και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιμένει να ακούσει τι έχουμε να σχολιάσουμε σχετικά με τα άρθρα αυτά πρωτού παρέμβουμε. Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμη είναι η απάντηση αλλά αυτά που μου μου λέτε ε, είναι πιο ικανοποιητικά σχετικά με το εκτιμώντας 31. Είναι το σημείο που νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς ε, να ε, παρεμβάλλει τις συλλογικές συμβάσεις και πρέπει να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μια σταθερή λύση αναλόγως του αν θα υπάρξει κανονισμός ή οδηγία. Γι' αυτό και θα θα παρακαλούσα στην περαιτέρω συζήτηση να δούμε αν το εκτιμώντας αυτό που είναι απλούστατα ε, η μισή πρόοδος δεν μας βοηθάει τόσο πολύ εφόσον είναι ε, προϋπόθεση. Εσείς θα κρίνετε να χρησιμοποιήσετε δηλαδή την προθεσμία για τις τροπολογίες και να προσθέσετε ένα άρθρο για τα εκτιμώντας με τα προβλήματα που σας απασχολούν. Και μετά ο εισηγητής θα συνθέσει. Ο κύριος Μπέκερ και μετά ο κύριος Κρίστιανσεν. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η εκτίμηση της οποίας χαίρει ο Τόμας Μαν αποδεικνύεται μία ακόμη φορά εδώ, παρόλο που έρχομαι από έναν διαφορετικό κόσμο που δεν είναι αυτονόητο, που υπάρχουν ορισμένα κροματικά κριτήρια και δεν υπάρχει ευρύ αλληλεγγύη ε, Παρόλα αυτά έχω δύο θέματα, δύο επιχειρήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν για ένα θέμα το οποίο θέλουμε να αποφασίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία. Καταρχήν, η λογική του κάθε λέγει ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα εάν 75% του κόστους είναι έξοδα προσωπικού. Είναι μια πολύ λεπτή τη λογική και ε, ε, πρέπει να απαντήσουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα σε ένα αεροδρόμιο και αυτό υποθάλπει τη θέση αυτής της εκθέσεως διότι οι ε, επιχειρήσεις και το προσωπικό από κοινού προώθησαν τη θέση αυτή. Όταν δηλαδή ε, το, η, επιχείρηση πιέζεται, δεν θα δεχθεί τα επιχειρήματά μας και αυτό νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν κάνουμε συζητήσεις προς τα έξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω, θα ήθελα να ξέρω, εάν είναι δυνατόν να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο και ένα ανώτατο επίπεδο για το βάρος μιας βαλίτσας. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα με την μεταφορά των αποσκευών θα έπρεπε να ορίσουμε ένα ανώτατο ποσό κιλών ε, αναβαλίτσα ή θα πρέπει να την σημαδεύουμε, να την επισημαίνουμε τη βαλίτσα, να βάζουμε κάτι που να λέει ότι η βαλίτσα είναι πιο βαριά, όταν την παίρνει δηλαδή το προσωπικό των αεροδρομίων. Βλέπω λοιπόν ότι η δημιουργικότητα τρέχει. Ο κύριος Μπενιό και μετά ο κύριος Ντεμπακέρ. Ε, κάτι πάρα πολύ σύντομο να σας αναφέρω. Όλη αυτή η συζήτηση είναι λίγο ακαδημαϊκού χαρακτήρα, γιατί πάρα πολλά έχουν ανοίξει τις υπηρεσίες εδάφους, τις έχουν απελευθερώσει και είναι πλήρως ελεύθερη, απελευθερωμένη, απορριθμισμένη αγορά και μόνο περί τραγωδίας και αναβαγή δεν πρόκειται. Μίλησαμε και με τις αεροπορικές εταιρείες και είναι πολύ ικανοποιημένε από τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Σε όλα αυτά τα κρατημέλη που ε, συνέβη αυτό. Επίση, έχω να σας πω ότι όπου και να καταλήξει αυτή η υπόθεση, πρέπει να εξασφαλίσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν την εθνική τους αρμοδιότητα και η απορρίθμιση να γίνεται σε κάθε κράτος με τον τρόπο που τους αρμόζει το καθένα. Αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί φοβάται ο κόσμος για το τι θα γίνει άμα ανοίξει η αγορά. Πάντως, μέχρι στιγμής η κατάληξη ιστορίας ήταν μια χαρά, οπότε δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται υπερβολικά τον Μπέκερ. Και εγώ να έρθω με αυτά που είπε ο φίλο Μπένιον. Καλή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, γιατί έτσι θα έχουμε βελτίωση τη κατάσταση εν γέννη και από κοινωνική πλευρά γιατί δεν θα γίνει μόνο, μόνο κοινωνικό ντάμιγκ δεν θα γίνει. Έχει γίνει πολύ σε πολλά αεροδρόμια χωρίς να έχουν επιδεινωθεί οι συνδικές εργασίες. Και αντίθετα, σε κάποια αεροδρόμια που υπάρχουν ακόμα περιοριστικοί όρια για το πόσες εταιρείε μπορούν να ε, διαχειρίζονται, ε, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο καλά. Άρα, τουλάχιστον ε, ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα. Στη χειρότερη περίπτωση. Και εδώ η Επιτροπή προσπαθεί και η κοινωνική προστασία να σταθμίσει και την απορρίθμιση της αγοράς. δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι υπάρχει ποιότητα υπηρεσιών. Θα πρέπει να γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού, θα πρέπει να προσέχουμε τα στάνταρ, τα ποιοτικά. Γι' αυτό σας λέω. Είναι καλά ζυγισμένη η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά ας μην τα ξεχνούμε. Και την κοινωνική διάσταση όταν συζητάμε το θέμα. Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ε, σας στέλνω τους χαιρετισμούς της Επιτροπής Μεταφορών επί του θέματος σχετικά με την κοινωνική διάσταση εάν κοιτάξουμε την παραγωγικότητα των εργαζομένων υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί ακριβείς και ε, κατανείμονται μέσα σε μία ημέρα ε, διότι τα αεροπλάνα δεν φτάνουν όλα μαζί υπάρχουν ώρες εχμής και ώρες μεγαλύτερης χαλαρότητος και βεβαίως στη μεγάλη εχμή μειώνεται η παραγωγικότητα αυτή τη στιγμή είναι στην ε, η παραγωγικότητα στη Φραγκφούρτη 70% και στο Skip Hall στο Άμστερνταμ 61%. Άρα ε, δεν ξέρω ε, ε, ποια είναι και η οικονομική προστιθέμενη αξία της παραγωγικότητας στα πλαίσια αυτά, αλλά οι κοινωνικές συνθήκες οι οποίες θα επιβαρύνουν τον εργαζόμενο είναι της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Μπορεί μετά από ένα χρόνο να μην υπάρχουν πλέον οι ίδιες προδιαγραφές εξού και θα πρέπει να ε, εξετάσουμε και το θέμα αυτό πρώτου αποφασίσουμε. Κύριε Χάντελ, θέλετε να δευτερολογήσετε. Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Μεταφορών. Μήπως γνωρίζει ε, ποια, πώς άλλαξαν οι συνθήκες ε, εργασίας ε, εις τα γερμανικά αεροδρόμια που μειώθηκαν μισθοί μέχρι 48% χωρίς συλλογικέ συμβάσεις. Οπότε σχετικά με το άρθρο 13α της BGB θα πρέπει να ξέρουμε εάν εξασφαλίζονται οι συνθήκες ε, ε, αμοιβή και εργασίας ε, των εργαζομένων διότι υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε μείωση των κοινωνικών παροχών και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ούτε η Επιτροπή Μεταφορών. Μην δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ματίας Γουτ, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Εγώ δεν έχω τη γερμανική εμπειρία στον κλάδο, αλλά υπάρχουν ε, τρία πράγματα που με ανησυχούν σε αυτήν την ε, νομοθεσία και χαίρομαι που η Επιτροπή μας συνεργάστηκε με την Επιτροπή Μεταφορών είναι φυσικά το θέμα της προστασίας των εργαζομένων αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων διότι η προστασία για τα κοινωνικ... τα στα πλαίσια του κοινωνικού δικαίου σε ένα περιβάλλον όπου ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστια πίεση με την απολευθέρωση της αγοράς, η διάρθρωση του κόστους, οι εταιρείε low cost οι οποίες μέσω της μείωσης αυτών των υπηρεσιών προσπαθούν να μειώσουν και τις δαπάνες τους αλλά και το θέμα της ασφάλειας διότι τα αεροδρόμια είναι χώροι όπου παίζονται ιδιαίτερα το, το θέμα της ασφάλειας και η πίεση αυτή η προσαπολευθέρωση θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των εγγύσεων σε αυτό τον τομέα. Υπάρχει όμως και κάτι πιο συγκεκριμένο που με ανησυχεί. Δηλαδή, όταν έχουμε αλλαγή operator, θέλουμε να ξέρουμε πώς τα κεκτημένα κοινωνικά δικαιώματα μεταφέρονται στον νέο λειτουργό, στον νέο operator. Υπάρχει ένα λόμπινγκ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Υπάρχει ένα τεράστιο λόμπινγκ το οποίο θα ασκηθεί και στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Μεταφορών. Λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά και αυτές, αυτή η πίεση που θα ασκηθεί Όταν πρόκειται για αλλαγή παρόχου υπηρεσίας ε, ε, στο, ε, στο έδαφος, θέλουν να πετύχουν να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του κοινωνικού κεκτημένου, όταν περνάμε δηλαδή από τον έναν πάροχο υπηρεσιών στον άλλον. Ο κύριος Ματίας Γουτ από την Κομισιόν. Πού είστε? Α, εκεί. Ωραία, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα επέμβω γερμανικά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την έκθεση διότι είναι μια πολύ εκτενής έκθεση και φαντάζομαι ότι ολόκληρη η πρόταση θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του πακέτου αεροδρομίων διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στον τομέα των αερομεταφορών. Ξέρουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες πιέζονται πάρα πολύ από την παγκοσμιοποίηση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μία μία μεταμόρφωση των αεροπορικών μεταφορών στην ε, ε, Ευρώπη κατόπιν της ε, παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό και πρέπει να επιζητήσουμε μία ισορροπία. Αυτό θέλουμε και να ε, βασιζόμαστε περισσότερο στα κοινωνικά δικαιώματα με μια προσεκτική και επιφυλακτική απελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί παρόλο που από το 1996 έχουν ήδη απελευθερωθεί πολλές και το βλέπετε στα καλύτερα αεροδρόμια ότι έχουμε τα καλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο στην Ευρώπη από πλευρά αγοράς καταστημάτων παραδείγματος χάρη. Μέχρι στιγμής λοιπόν θέλω να σας υπενθυμίσω έναν αριθμό. Αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για αεροδρόμια με πάνω από πέντε ε, ε, ε, 5 εκατομμύρια επιβάτες έχουμε πάνω από 60 αεροδρόμια που είναι αντικείμενα αυτό ε, των προτάσεων 41, 19 ε, δεν έχουν ακόμη ανοίξει και 41 έχουν ήδη απελευθερωθεί θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν καλύτερες ποιοτικέ υπηρεσίες κανόνες ε, επίσης για την ανάληψη του προσωπικού σε περίπτωση αναμορφώσεων και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Απ' την άλλη πλευρά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε την κατεύθυνση η οποία υιοθετήθηκε σε ορισμένα κράτη-μέλη, δηλαδή συγχωνεύσεις. Θέλουμε να υπάρχει ένα ισορροπημένο κοινωνικό πακέτο το οποίο να προσφερθεί και συγχρόνως να πρέπει να οδηγήσει σε μία μείωση των αεροδρομίων και να δούμε εάν στην Ευρώπη ε, ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε τα μεγαλύτερα κομβικά αεροδρόμια για, την, για τις παγκόσμιες αερομεταφορές και να μην είμαστε απλούστατα στα αεροδρόμια σε εξωτερικά σκέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το hub, το κομβικό αεροδρόμιο να βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε πολύ έντονα στην Ευρώπη, αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας προτείνω να σκεφτείτε είναι ότι θα χρειαστούμε συγκεκριμένους κανόνες για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν υπάρχουν. Ε, αλλά μέχρι στιγμής ήδη υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου προέχουν συνθήκες ε, ε, όπου υπάρχουν 5, 6, 7 εταιρείες ε, εξυπηρετήσεως για το, τις υπηρεσίες εδάφους και με αυτό θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Χαίρομαι ότι εσείς υγείστε της διεκπαιρεώσεως αυτού του θέματος και χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι στη συζήτηση μεταξύ Επιτροπής Μεταφορών και Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών θα βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ σας. Φαντάζομαι κύριε εισηγητά ότι θα μιλήσει γερμανικά. Ναι, Ξέρω ότι στη συνέχεια έχουμε ψηφοφορίες, οπότε καταρχήν θα πω ελάχιστα. Ε, ευχαριστώ για όλα τα καλά σχόλια που είναι μία ένδειξη ότι έχουμε μία έκθεση ε, στην οποία ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αντικατοπτρίζονται οι ιδέες μας. Επίσης όσον αφορά τις μειώσεις μισθών συμφωνώ με την γενική άποψη ότι εγώ δεν μιλάω μόνο για τα αεροδρόμια της χώρας μου, μιλάω και για άλλες χώρες. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι πάροχοι εκεί και ενδεχομένως δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν οι ισχύσεις συνθήκες. Αυτό που θεωρώ επίσης σημαντικό γιατί με ε, τηγόρησαν ότι ε, ε, ο εισηγητής είναι από μια συγκεκριμένη χώρα, πολύ παρενέβησα στη γλώσσα μου, γερμανικά δηλαδή, αλλά δεν έχουμε εμπειρίες μόνο από τη Γερμανία, έχουμε και από την Ελλάδα και από τον Μπρίστολ και από άλλες χώρες όπου υπάρχουν διαφορετικές διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές δυνατότητες συνδέσεως, αλλά πρόκειται για χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένας βασικός τομέας. Για την μετεκπαίδευση, να υπάρχουν ενιαία πρότυπα εκπαιδεύσεως. βέβαια σε δύο μέρες δεν τα μαθαίνει κανείς όλα. Εμείς ε, θέλουμε να υπάρχει ε, κρατικός έλεγχος των εξετάσεων για προσωπικό αεροδρομίων για να υπάρχουν ασφαλείς ε, κατευθυντήριες γραμμές, ε, σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και όλα αυτά βέβαια κοστίζουν και οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αμείβονται ικανοποιητικά. Μας ε, είπες ότι είναι πολύ βασική παράγραφος 50 και αυτό θα είναι σημαντικό και στην Επιτροπή μεταφορά. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μία ενιαία αντιμετώπιση. Είμαστε ε, συνδεδεμένοι στην προσπάθεια αυτή με την Επιτροπή Μεταφορών. Τόμας Χέντελ, ε, ευχαρίστως ε, βλέπω η Γκούε να στηρίζει τους χριστιανοδημοκράτες. Είπες ότι υπάρχουν σημεία που θέλουν περαιτέρω σκέψη, το σημείωσα και και είπες ότι ορισμένα περίφθησαν πολύ σωστά και συμφωνώ διότι τα αεροδρόμια κατέληξαν σε κοινέ αποφάσεις μεταξύ ε, εργοδοτών και εργαζομένων πολλές φορές υποπίεση αλλά ε, αυτά έγιναν για να μπορέσουν να ε, επιβιώσουν αν μπορούσαν τα αεροπλάνα να κινηθούν χωρίς ε, βοήθεια προσωπικού και των υπηρεσιών εδάφου τότε ενδεχομένω θα μειωνόταν το κόστο, κόστος αλλά πολύ σωστά είπες ότι πρέπει να ξέρει κανείς για κάθε αποσκευή που βρίσκεται, τι βάρος έχει, πώς διακινείται και θα χρειαστεί στην Επιτροπή μας και λίγη δημιουργικότητα. Ε, κύριε Μπέγγελ, ε, γνωρίζω το βρίσκο Μπρίστολ και το Χήθρο. Όποιος έχει πάει στο Λονδίνο στο Χήθρο ξέρει ότι υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις παρόλο που υπάρχουν πολλοί πάροχοι. Ε, υπολογίζω ότι έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα καθυστέρηση εκ προημίου ενώ αλλού έχουμε το πολύ 10 λεπτά. Ε, βεβαίως ε, πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε όλες τις πτυχές, τόσο Σέγγεν, όλα, όλα αυτά κοστίζουν χρήματα ε, ευχαριστώ όμως για τη συζήτηση κυρία Πρόεδρε. Ε, όπως είπες, ε, ελαρζεμό opérateur. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρχει μία στενή συνεργασία και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσει σοβαρά τις επιφυλάξιμες. Εμείς θέλουμε ανταγωνισμό αλλά να είναι δίκαιος, να υπάρχουν σωστές συνθήκες. Οι άνθρωποι να αμείβονται ικανοποιητικά και λογικά. Και προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε περαιτέρω μεταξύ μας και σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ αγαπητέ εισηγητή. Λοιπόν, 27 Ιουνίου στις 5 ε, η δημιουργικότητά σας είναι ελεύθερη μέχρι τότε. Σας ε, παρακαλώ να αποφύγουμε να έχουμε χίλιες τροπολογίες για μια γνωμοδότηση. Αυτή, αυτή είναι πόθη, ευσεβής πόθη της ε, Προέδρου βέβαια. Πάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχουμε μία σημαντική ψηφοφορία, πρόκειται για την πρώτη νομική βάση για την οποία θα εκφραστεί η Επιτροπή μας εν ώψη της επόμενης διαπραγμάτευσης των δημοσιονομικών προπτικών. Και έχουμε 120 συμβιβαστικές τροπολογίες. Όλοι έχετε την κάρτα σας, εγώ δεν την έχω. σχόλιο του κυρίου Μαν εκτός μικροφώνου και απαντάει πρόεδρος, εγώ θα πήγαινα να, τη, να την ψάξω αλλά θα καθυστερούσα. Άρθρο 1, παράγραφος 1. Συμβιβασμός σε σε. Τμήμα ενός μπλοκ 1. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός DD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Β το αρχικό κείμενο της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το άρθρο 2 Παράγραφος 1 δέλτα, το ε ε υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2 παράγραφος 1 μετά από το σημείο D ένα νέο σημείο βάση του συμβιβασμού FF. Υποστηρίζεται από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο D πάντα νέο σημείο με έναν συμβιβασμό πι, πι, πι. Που δεν είναι τα αρχικά παρτεναριά public Πριβέ. Λοιπόν, πι, πι, πι λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο δέλτα β, ΔΜΠ, συμβιβασμός ΖΖ. Υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγικό τμήμα ψηφίζουμε ένα νέο μπλοκ, ε, μπλοκ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο α συμβιβασμός ή ή. Τέσσερις ομάδες το παρουσιάζουν υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο Β, συμβιβασμός ζ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο σ. συμβιβασμός κ. Κακά λέει η πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο γ, σε δηλαδή α λ λ συμβιβασμός μπλοκ 2 το ψηφίσαμε άρθρο 3 παράγραφος 2 μπλοκ 3 υπέρ υποστηρίζεται από τέσσερις ομάδες δεν πρέπει να διστάζετε να το υπερψηφίσετε λοιπόν. Υπέρ. Μπλοκ 3, μπλοκ 3. Είναι ο συμβιβασμό M, M, X, X, H, H, e, e, κλπ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4. Παράγραφος 1 σημείο α. Συμβιβασμός εν εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο β. Συμβιβασμός ο, ο, ο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο γ. Συμβιβασμός π, π. κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο σε έχουμε την τροπολογία 234 του κυρίου Κοσλόφσκι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 4 παράγραφος 1 μετά από το σημείο σε Έχουμε ένα νέο σημείο με την τροπολογία 235 της κυρίας Τζίμερ, του κυρίου Χέντελ και Λεγιαρίκ. Έχουμε μια προφορική τροπολογία του εισηγητή, συμφωνείτε με την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε τη 235, υπέρ, κατά, άποχες. Εγκρίνεται άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο D, δέλτα. Κι κι Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1, μετά από το σημείο D, Επιτροπή Γυναικών, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται, εισηγητής είναι υπέρ. Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο C, συμβιβασμός RR. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 1 μετά από το σημείο ε ένας συμβιβασμός S, S από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. μετά από το σημείο 1 έχουμε τον συμβιβασμό TT που υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 2 εισαγωγή Τροπολογία 41 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο α συμβιβασμός βέβαια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο β συμβιβασμός βέβαια από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4. Με νέο άρθρο 4. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, όχι. Άρθρο 5 παράγραφος 1. Συμβιβασμός Y, Y, Y, Υπερκαταποχές. Εγκρίνεται άρθρο 5 παράγραφος 2. Υπό παράγραφο 1 εισαγωγικό τμήμα συμβιβαστική ZZ υπέρ κατά εγκρίνεται άρθρο 5 παράγραφο 2 υπό παράγραφο 1 σημείο α συμβιβαστική ΑΑΑ παρουσιάζεται από πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, σημείο Β, συμβιβασμός BBB, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, σημείο C, το πρωτότυπο της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Άρθρο 5, παράγραφος 2, παράγραφος 2, συμβιβαστική ΣΣΕ, τρεις ομάδες υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Η 50 αποσύρθηκε, άρθρο 5, μετά από την παράγραφο 2. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τον συμβιβασμό DDD, τον ψηφίσαμε ήδη. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, μετά την παράγραφο 2, νέα παράγραφος με τον συμβιβασμό εεε ε ε, υπερκαταποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5 παράγραφος 3 συμβιβασμός FFF υπερκαταποχές εγκρίνεται. Σημείο 6. Παράγραφος 1, σημείο 1, σημείο α. ΖΖΖ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο 1, σημείο β, 53 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο 1, σημείο σ, συμβιβασμός ας, ας, ας, h, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημειώνε μετά από το σημείο D η 55 του εισηγητή κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 1 μετά από το σημείο D 276 της κυρία, των κυρίων Ντελή και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 277 κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 1, σημείο 1, ο συμβιβασμός 3 ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 2 σημείο β, τροπολογία διαγραφής. Και ψηφίζουμε μαζί την 58 και 280 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο 2 κλπ. του κυρίου Μπουλό για να διαγραφεί... Α, αποσύρθηκε αυτή η τροπολογία, συγγνώμη. Όπως και η 282 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό ZZZ που έχουν παρουσιάσει τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο 2, σημείο D, 284 του κυρίου Μπουλό με προφορική τροπολογία, δεν υπάρχει αντίρρηση, ψηφίζουμε την 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο 2, μετά από το σημείο ΜΙΟΕΦ της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 287 της κυρίας Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές αποχές εγκρίνεται 288 της κυρίας Στάιρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 3 σημείο β 3 κ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 3 μετά από το σημείο B συμβιβαστική τροπολογία 3 λάμδα 4 ομάδες υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 3 μετά από το σημείο Β 62 του συγητή υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 3 σημείο C σημείο γάνομα δηλαδή 19 της Ήτρε υπερ κατά αποχές. Θέλετε να το παληθεύσουμε. Να αλλάξουμε το ρυθμό της ψηφοφορίας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 23 υπέρ 17 κατά. Εγκρίνεται. Δεν καταψηφίζουμε τίποτα σήμερα το πρωί. 26 συμβατή της Ρέγγι υπέρ η κυρία Στάρμπεκ. Έχουμε μία προφορική τροπολογία η οποία λέγει... Ε, organization in all fields. Euh, le texte dit organisation de travailleurs, de groupes Οργάνωση των ομάδων των εργαζομένων και ο εισηγητής προτείνει διεθνικές οργανώσεις εργαζομένων. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 26 της ΡΕΓΚΙ όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο 3, σημείο δέλτα, συμβιβαστική τροπολογία 3 μη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 συσυγήτρες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 27 της Ρέγγι θα έχουμε την ίδια προφορική τροπολογία, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε την παράγραφο 27 της Ρέγγι υπέρ κατά 27 ούτως τροποποιημένη εγκρίνεται. Συμβιβασμός Τρία νη από 4 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 4 σημείο β Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο 5. 3 όμικρον. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7, συμβιβασμός 3Q. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3R. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8, 67 της ε, εισηγήτρας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8 παράγραφος 2, 315 των κυρίων Ντελή και υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 8 παράγραφος 2, νέα παράγραφος, 32 της Ρέγγι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 9 παράγραφος 1, 69 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε το 69. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 22-19. Εγκρίνεται. Άρθρο 10 παράγραφος 1, συμβιβασμός 3S. Τέσσερις ομάδες το παρουσιάζουν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 10 παράγραφος 1 καινούριο, 70 της εισηγήτρες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 της εισηγήτρες υπέρ, Κατά. Υπέρ της 71. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 11 παράγραφος 2. 10 του ελέγχου του προπολογισμού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 ελέγχου προπολογισμού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 ελέγχου προπολογισμού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 13 συμβιβασμό ταφ ταφ ταφ ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 14 παράγραφος 1 γιου γιου γιου γιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 14 μετά από την παράγραφο 1 73 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 74 πάλι της εισηγήτριας εγκρίνεται. Άρθρο 14 παραγραφός 2, συμβιβασμός 3 βιτ, Β. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τίτλος 2, 75 της εισηγήτρες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 14 νέο, συμβιβαστική 3 W, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15, παραγραφός 1, αγωγικό τμήμα 3, χ, 4 ομάδες υπερκατάποχες εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο α, 3 ε, υπερ κατά εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο β, 3 ζ, 4 ομάδες υπερ κατά εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 1, μετά από το σημείο Β ήταν νέο σημείο. Συμβιβασμός 4 σε 4 μαζί κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο σε 4α υπέρ 5 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο Δ, συμβιβασμός 4β, Τέσσερις ομάδες. Η υπερκαταποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15 παράγραφος 2 σημείο β. Χωριστή ψηφοφορία στο πρωτότυπο της Κομισιόν. Α, είπα 15, όχι, όχι, πάμε, δεν είναι σωστό αυτό, 16, 16 είναι. Παράγραφος 2, σημείο Β. Το πρωτότυπο τη Κομισιόν υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Άρθρο 16, παράγραφος 2, σημείο σε. 4 ε. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Άρθρο 16, παράγραφος 2, σημείο ε, 4D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 16, παράγραφος 3, τροπολογία 84 της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να το παληθεύσουμε, ας επαληθεύσουμε, νομίζω ότι πέρασε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 22... 17 μια αποχή εγκρίνεται. Άρθρο 16 παράγραφος 4 συμβιβασμός 4F που παρουσίασαν τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 17 Ψηφίζουμε. Α, το άρθρο 17 δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε, λέει η Πρόεδρος. Μετά από το άρθρο 19 πρέπει να ψηφίσουμε το 4G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 20, παράγραφος 1, σημείο α, 4K, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 20, σημείο 1, παράγραφος 1, σημείο β, τα 4 λάμδα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 20, παράγραφος 1, σημείο β, νέο, συμβιβασμός 4, νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 20 μετά το νέα παράγραφος. Τα τέσσερα μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από το άρθρο 20, ένα νέο άρθρο 355 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο άρθρο 21 παράγραφος 2 το εισαγωγικό τμήμα. Την 94 ε, της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το πρωτότυπο κείμενο της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 21 παράγραφος 2 σημείο γάμα Συμβιβασμός 4 όμικρον που έχουν παρουσιάσει τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 21, παράγραφος 2, νέο, 98 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 21α νέο συμβιβασμός 4π που έχουν παρουσιάσει τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 21 παράγραφος 1 εισαγωγικό τμήμα συμβιβασμός 4 ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 22 παράγραφος 1 σημείο 1 σημείο α τα 4 Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 22 παράγραφος 1 σημείο 1 νέο σημείο συμβιβαστική 4 ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 22 παράγραφος 1 μετά από το σημείο 2 νέο σημείο τροπολογία 365 του κ. Μπουλόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άρθρο 22, παράγραφος 1, σημείο 2, νέο, 4 σίγμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 22, παράγραφος 1, σημείο 3, καταπίπτει. Άρθρο 22, παράγραφος 1, νέα, συμβιβασμός όμικρον. Μα τι θέλει εδώ στη μέση αυτό, λέει η πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ της ο. Εγκρίνεται. Άρθρο 22, παράγραφος 1, 4, γιου. Τέσσερις ομάδες παρουσιάζουν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 23, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα, το πρωτότυπο της Κομισιόν, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 23, παράγραφος 1, σημείο 1, τα 4 β, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 23, παράγραφος 1 σημείο β, το πρωτότυπο της Κομισιόν υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρθρο 23 μετά την παράγραφο 1, νέα παράγραφο συμβιβασμός 4W υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρθρο 23, παράγραφος 2, συμβιβασμός 4χ, υπερ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 23, παράγραφος 3, συμβιβασμός 3y, 4y, ε, ε, συγγνώμη, υπερ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 24, συμβιβασμός ζήτα, υπερ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα κάνουμε ένα upgrade των συμβιβασμών. Έχουμε μία συμβιβαστική 5α. Υπερκαταποχές εγκρίνεται. Άρθρο 25 παράγραφος 1 συμβιβασμός 5β. Υπερκαταποχές εγκρίνεται άρθρο 25 παράγραφος 1 μετά την παράγραφο 1. 5 σε υπερα κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 25 παράγραφος 2, 5D, υπερ... Α, καλύφθηκε, καλύφθηκε, συγγνώμη, συγγνώμη. Ψηφίζουμε, άρθρο 25 παράγραφος 3, την παράγραφο 23 της Επιτροπής Προλογισμών υπερ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 25 παράγραφος 4 και αυτή έχει καλυφθεί. Άρθρο 26 παράγραφος 1 5G υπέρ αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 26 παράγραφος 2 τα 5H υπερκάτα αποχές εγκρίνεται. Όχι 25, αφού 100. Άρθρο 25. 2. 125 της Όχι μετά. είναι υπέρ του 125 της εισηγήτριας. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Φτάνουμε στον τίτλο που έχει καλυφθεί και ήδη έχουμε φτάσει στις ιδεολογικές παραγράφους. για τις αιτιολογικές παραγράφους στην παριθμόν 3 ψηφίζουμε το τη συμβαστική σε πέντε πολιτικών παρατάξεων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Συμβαστική δε είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε που θα επανενταχθεί στο κείμενο ως νέο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά το 4, παράγραφος 2, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά το 4, τροπολογία 136 της κυρίας Τσίμερ, κυρία Χέντελ, με προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια. Υπάρχει κάποια ένσταση, όχι από ό,τι φαίνεται, επομένως ψηφίζουμε το 136. Τσίμερ Χέντελ Πιπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά έχουμε το 137 της ηγετρίας και της κυρίας Ρέγνερ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με το 4 παράγραφος 2, την Επιτροπή Γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ, δύο Επιτροπή Γυναικών. Παράγραφος 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στο 5 έχουμε το F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ε, κατόπιν ε, έχουμε την επόμενη που κατά η συγκύτρια υπέρ κατά εποχές και απορρίπτωται. Παλήθευση. Ψηφίζουν. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 21 υπέρ, 18 κατά και μία εποχή. Έχετε δίκιο, διότι εγκρίνεται. Πράβος 2. Ελέγχου προπολογισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 5. Παραγραφός 3. Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην ε, αιτιολογική 6 έχουμε το ζ από 6 εποχές ομάδες υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 7 συμβαστική H, H, ο τέσσερις πρωτιοσμάδες υπερκατά αποχές εγκρίνεται για την ιδεολογική 8 Γιώτα. Πέντε πολιτικέ ομάδε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Μετά το 8. Παράγραφος 5. Επιτροπή γυναικών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Από την Περιφερειακή Επιτροπή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. J. G. Τέσσερις πολιτικές ομάδες. αιτιολογική 10, κάπα, 4 πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 11, συμβαστική L, 4 πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 12, 157. Από τρία μέλη της Γκουέι και ζητούν κάποια απαλληλήφη, Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. αιτιολογική 12. Τώρα τη συμβαστική M, τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και είμαστε τώρα στην ε, τροπολογία 10 της εισηγήτριας υπέρ κατά. Αποχές. Επαλήθευση για το 10. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 17. 23. Μηδέν αποχές. 16 λέει η συσκευή. Επομένως απορριβέται και. Πάμε τώρα στο 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 συγκίτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 ζητείται απαλληφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. Αιτιολογική 14. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Δεκαπέντε συμβαστική π. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Q υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Δεκαεπτά. Το R. Τέσσερις πολιτικές ομάδες υπερκατά αποχές. Εγκρίνεται. το 17. Έχουμε το 178. τέλει, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και μετά το 17 έχουμε το 179. τέλει. Εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Εδώ μέχρι εκεί που λέει ε, επιδοτήσεις ε, στην απασχόληση και σε, και στην ασφάλιση μέχρι εκεί ψηφίζουμε, πρώτο τμήμα ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 21-19. Εγκρίνεται το πρώτο μέρος. Και τώρα το δεύτερο τμήμα σε παρένθεση να προσθεθούν αυτά τα οποία αφαιρέσαμε στο πρώτο ήμιση. Περ, κατά, αποχές. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτωται. Και τώρα, μετά το 17, πάμε στο 180. Ντέλη πάλι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. W. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μετά το 18 Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 18 τροπολογία 184 Ντέλη και Σρέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 18 ψηφίζουμε το 19. Αιτιολογική 19, συμβαστική χ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Τι ηγητρίας. Υπέρ. Αποχές ε, και εγκρίνεται μετά το 19 187. Τρεμόσα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει επαλήθευση. Πέρασε. 21 υπέρ 17 κατά που είναι εγκρίνεται εκτιμώντας 20 γλωσσική τροπολογία μετά από το εκτιμώντας 20-22 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 ψηφίζουμε το πρωτότυπο της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά από το 22 ψηφίζουμε την 7 της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ κατά άποχες. Επαληθεύουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ 21 κατά Απορρίπτεται. Συμβιβασμός Συμβιβασμό Τέσσερις ομάδες το ψηφίσαμε στον μπλοκ 3 αυτό. για το νομοθετικό ψήφισμα. Κυρία Στάνιο. Αν κατάλαβα καλά, ε, το σημείο 97 δεν έχει ψηφιστεί. L'amendement 97. Η τροπολογία 97 θα κατέπευτε άμα θα παίρναγε 357 ε, η οποία θα κατέπευτε με τη σειρά της και λοιπά οπότε δεν καταλαβαίνω πώς λοιπόν παράγραφος 1 της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 1, παράγραφος 2 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συνολικά το κείμενο δια ηλεκτρονικής οδού. Αρχίζει η ψηφοφορία. Vous voulez pas de vote électronique? Δεν θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μα ναι, μα ναι, λέει η πρόεδρος. Mm. Ψήφισατε όλοι. Εκτάκτος πως 36 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Pour ce brillant succès για αυτήν τη λαμπρή επιτυχία. Να σας πω ότι κρατήσαμε μόνο έξι μικροσημεία της, ε, μικροτμήματα της Κομισιόν. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν είναι εδώ. Και μεταξύ αυτών των έξι μικρών τμήματων τα περισσότερα αφορούν στα εισαγωγικά του κειμένου. Καταλαβαίνετε την ε, σκληρότητα των διαπραγματεύσεων της και της διαπραγματευτικής διαδικασίας και το βάχρος του έργου των, των διαπραγματευτών. Εμείς ευχαριστούμε και για τον αριθμό των τροπολογιών την εισηγήτρια και θέλω να ευχαριστήσω και τα δύο μέλη της γραμματείας που συνεργάστηκαν στενά για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν όλη τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Και, δεν υπήρξε, και είχαμε μηδέν λάθος στην όλη τη διαδικασία. ευχαριστώ και τον Σκιώδη συγητή. Τώρα πάμε στην έκτακτη διαδικασία να σας διαβάσω κάτι. Πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτήν την ψηφοφορία ξεκινάμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για μια πιθανή συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Σύμφωνα με το άρθρο 70 και την παράγραφο 21 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Προτείνω, αν συμφωνείτε βέβαια, σύμφωνα με τις διατάξεις των κειμένων που διέπουν τις εργασίες μας, η διαπραγματευτική ομάδα να αποτελείται από τη μία μεριά της υποφαινόμενης, της εισηγήτριας και των σκιωδών εισηγητών. Αυτό σημαίνει ότι οι υποφαινόμενοι, η κυρία Στάριοκ, ο κύριος Μπούλα, η κυρία Χάρκιν, η κυρία Ελίζαμπετ Σρέτερ, η κυρία Καρή Μαντελή. Μια, μια από τις δύο, ε, όχι και οι δύο στον τρίλογο η Γκαμπριέλα Τζίμερ και Ανδρέα Μακεντήρ. Η διαπραγματευτική εντολή αποτελείται από την έκθεση την οποία εγκρίναμε με τους όρους που γνωρίζετε και ο πρώτος τρίλογος με το Συμβούλιο και την Κομισιόν προβλέπεται στις 10 Ιουλίου 10 Ιουλίου τώρα φέτος στις 18 και και θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις της διαπραγμάτευσης. Τα σημεία 22 και 23 έχουν αναβληθεί. Πάμε στο σημείο 24. Γνωμοδότηση της κυρίας Γιώτοβα για τι συνθήκε εργασία των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών, για την Επιτροπή Γυναικών επί τη ουσία. Μου λένε ότι στον κατάλογο ψηφοφορία υπάρχουν δύο αλλαγέ. Προφορική τροπολογία στο 11. Δεν αφορά την 11, αλλά αφορά την 27. Και η τροπολογία 12 έχει αποσυρθεί. Λοιπόν, παράγραφος 1, συνδυασμός α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 1, τροπολογία 10 τη της κυρίας Ζούμπερ και του κυρίου Λεγιαρίκ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το calls on the commission may work such shifts. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα βεβαίως και μπορεί να ψηφιστεί. Το δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 1, τροπολογία 11 της κυρίας Κλιβέτη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός, ε, παράγραφος 2 συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 κοχμερίν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 ε, Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 Πουπάκης καταπίπτει. 19 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 συμβιβασμό σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 συμβιβασμός δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 Κορνέλισεν με προφορική τροπολογία που ανέφερα προηγουμένως που παρουσίασε το ΕΛΚ και που αφορά στην αντικατάσταση calls on the με encourage αντί καλή ενθαρρύνει. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ψηφίζουμε την 27 όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 5 ψηφίζουμε τον συμβιβασμό ε, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 34 του κυρίου Μπερμάιερ, υπέρ κατά αποχές, αποχές. Θα το επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 34. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 16 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Θα... Άκουσα, άκουσα, λέει ο πρόεδρος, άκουσα. Αμπά. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω αυτό. 32 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 κλιμπέτη εγκρίνεται. Διορθώσαμε το λάθος μου. Πάμε στην 35 της κυρίας Κίνγκα Γκέντς. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 6. Unblock. Unblock όλα τα υπόλοιπα Ωραία. Όλοι συμφωνείτε για την παράγραφο 6 κλπ. Σύμφωνοι, ωραία, υπέρ. Κατά αποχές ψηφίζουμε συνολικά την ε, γνωμοδότηση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ 2 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πάμε στο σημείο 18 που δεν εξετάσαμε χθες. qui nous conduit à donner la parole. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ. Για σιωπή, λέει ο πρόεδρος. Για την γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Γεωργίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Αλάσσιες Υποθέσεις και την Αλία. Έχετε το λόγο κυρία η συγγήτρια για να μας παρουσιάσετε τις 73 τροπολογίες τις οποίες εισάγατε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ συνολικά στο τι θα συζητηθεί. Με την μεταρρύθμιση του Ταμείου για τις Ελλάδες Υποθέσεις και την Αλία θέλουμε να απλουστεύσουμε τις, ε, την νομοθεσία και να προσεγγίσουμε τις ε, αρχές της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης ε, θαλάσσης πολιτικής. Μέχρι το 2020 θα πρέπει να εφαρμοστεί και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους στρατηγικής 2020 μέσα από τρεις πρωτοβουλίες. Πρώτη η Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί σωστά τους ελευτικούς πόρους, μετά η καινοτομία και τρίτο νέες ειδικότητε και θέσεις απασχόλησης. Για τη δική μας γνωμοδότηση θα πρέπει να τονίσουμε πλευρές που θεωρούμε απαραίτητες για να βελτιστοποιήσουμε την απασχόληση, να είναι δηλαδή απασχόληση ποιότητα, να καταπολεμάει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, να ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και την χωροταξική ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε ε, εδώ ειδικά τους ε, αλίες, ε, τους, τους τους βιοτέχνες πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας την βιοτεχνική αλληλεία διότι και απασχόληση δημιουργεί και λιγότερες ζημιές κάνει στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για να αποφύγουμε την εξαφάνιση παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από τον αλλιευτικό τομέα θα πρέπει να εγγυθούμε αηφόρες δραστηριότητες της αλληλείας, μακροπρόθεσμα Πρέπει όμως να προωθήσουμε και τη διαφοροποίηση προς άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Πολλές φορές οι αλλοίς δεν εργάζονται ορισμένες ε, περιόδους και πρέπει να τους βρούμε μία λύση. Χρειάζεται κατάρτιση του αλλιέα, της οικογένειάς του και κυρίως των γυναικών που εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση. Η κατάρτιση θα πρέπει να είναι και αρχική αλλά και, μόνιμη, και βασική αλλά και μόνιμη. Ε, ε, θέλουμε επίσης να, επηρε, να ε, επηρεάσουμε την υγιεινή και την ασφάλεια εργασίας των εργαζομένων των κλάδων που είναι πολλές φορές τσαπατσούλικοι. για το θέμα της ασφάλειας, πέρα από το θέμα της ασφάλειας θέλουμε να επεκτείνουμε τον κοινωνικό διάλογο σε όλους τους κλάδους που καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών αλλιέων, τους οποίους συνήθως δεν τους λαμβάνουμε υπόψη και των οποίων η γνώμη θα πρέπει να εξαρθεί. Ε, Επίση θα πρέπει να, να συμπεριλάβουμε και την κοινωνική καινοτομία για να βρούμε νέες λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Αυτά πολύ σύντομα ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία βασίζουμε τις τροπολογίες μας. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμεί ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Σέρκας. Και ο κύριο Κρίστινσεν που θα είναι ο σχεδόν και εγώ ακούσαμε και τη την έκθεση της κυρίας Λόπη Φοντανία και συμφωνούμε 100% μαζί της με όλα όσα πριν από λίγο μας εξήγησε και το μόνο θέμα το οποίο πρέπει να σας πούμε είναι το εξή. Οι σοσιαλιστές επίσης προβληματιζόμαστε για το ότι υπάρχει εδώ αυτό το θέμα των γενεών, των, των, των, της γιατί όπω και με τη γεωργία θα πρέπει κάτι να κάνουμε όσον αφορά αυτέ τι απειλέ που επικρέμανται όσον αφορά την αηφορία, τη βιωσιμότητα και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει επίσης και με τους νέους φιλείς. Ε, πάντως δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Ε, συμφωνούμε με την εισηγητρία και όπως είπα και προηγουμένως. Ε, Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και συγχαρητήρια στην εισηγητρία για το έργο της. Ο επόμενος. Thank you, Madam President. Uh, just two points from the original text. Δύο τι να θέλουμε να πούμε, ο κ. Ε, σε σχέση με το αρχικό κείμενο στο τέλος. Στο τέλος ε, ανέφερε για την υποστήριξη των κοινοτήτων των Ελλήνων. Μα είναι αυτοσυντηρούμενοι, διότι ε, ανέκαθεν ψαρεύουν, γυρίζουν και οι κοινότητες τους, όσοι επιτοπλίστων δείτε το χαρτί της Ευρώπης, είναι μάλλον μικρές Υπάρχουν βέβαια και μεγάλες, αλλά οι περισσότερες είναι μικρές, μικροί λιμένες. Και οι περισσότεροι εξαρτώνται εκεί από την αλληλεία. Βεβαίω και αυτό ε, δημιουργεί τουρισμό, οπότε το σύνολο ε, ε, εξαρτάται από την αλληλεία και μέσα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι από νομοτικής πλευράς η υποστήριξη, η βοήθεια. Οπότε, ξαναγυρίζουμε τώρα στην αρχή του εγγράφου και η εν λόγω πρωτοβουλία μας λέει για την βοήθεια προς την κοινή αληθή πολιτική, η οποία όμως είναι ένα ναυάγιο, μια τραγωδία από το 1973 που ξεκίνησε. Έχουμε μείωση και μείωση των αληθικών πόρων. Δεν υπάρχουν πια ψάρια σε ορισμένε περιοχές και γι' αυτό ευθύνεται η πολιτική αυτή με τις απορρίψεις που πετάνε ε, λόγω αυτού του γελίου στήματο των προστώσεων πετάνε τόσο και τόσα ψάρια που έχουν ήδη αλλιεύσει νεκρά. Όμως, ας ξανακάνουμε την αλληλεία αυτή που πάντα ήταν. Ο καθένας να ψαρεύει στα, ε, στα χωρικά ύδατα, ο καθένας να προσέχει τους ελευτικούς του πόρους και έτσι η δραστηριότητά τους να πηγαίνει από τη μία γενιά στην άλλη. Και αν σας πω για δύο χώρες υπάρχουν στην στην Ευρώπη, Νορβηγία και Ισλανδία, που εξαρτώνται από την Αλία και ούτε μία ούτε οι άλλοι βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στις δύο περιπτώσεις ε, δεν έχουν προσχωρήσει στην αλληλευτική πολιτική, έχουν τη δική τους νομοθεσία. Οπότε εκεί οι, οι αλληλευτικοί πόροι και οι κοινότητες θα πάνε μια χαρά. Στην αρχή του ενός έτους είπε η Νορβηγία ότι αυξήθηκαν οι αλληλευτικοί της πόροι και κυρίως οι γόνοι. Πάνε πάρα πολύ καλά και ένα σωρό ε, είδη γεννούν και πολλοπλησιάζονται όπως πρέπει. Στην Ισλανδία επίσης ε, έχουν ε, απαγορευτεί οι απορρίψεις δε, στο δε Ηνωμένο Βασίλειο πιάνουμε πάρα πολύ λίγα ψάρια. Συνήθως ε, κάνουμε εισαγωγές από την Ισλανδία. Αυτοί επομένως ε, φρόντισαν τα χωρικά τους ε, ύδατα και τα πήραν μια χαρά και βρίσκονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να απαλλαγούμε από την κοινή αλληλευτική πολιτική και να σταματήσει αυτή η τραγική πρακτική του να πετώνται τα νεκρά ψάρια πίσω στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Λάμπετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, νομίζω ότι περισσότεροι εδώ ανησυχούμε για την κοινή ελευθερική πολιτική και για τι απορρίψει, αλλά νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν αλλαγέ στα χωρικά μα ε, ύδατα, αλλαγή στη θερμοκρασία, αλλαγή στο κλίμα κλπ. Και έχουμε ένα σωρό προβλήματα τα οποία έχουν πλήξει τις μικρές ελευτικές ε, παρακτής κοινότητες, όπως είπε και η συγγήτρια. Οπότε, όταν φτάνει η ώρα να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τι θα γίνει μέχρι το 2020, το θέμα της ε, βοήθειας αυτών των κοινοτήτων είναι πάρα πολύ άμεσο και νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογη αυτή η έκθεση που με τώρα συζητούμε. Φύγει όλα αυτά τα ζητήματα, ε, αυτά που μας τα εξήγησε η κυρία Φοντανιέ τη διαδοχή που γενιά σε γενιά, που είπε και ο κύριο Θέρκας, την κατάρτιση και όλα αυτά. Επομένω νομίζω ότι ε, έχει λάβει τη σωστή κατεύθυνση η υπόθεση με αυτή την έκθεση. Δεν βλέπω άλλον συνάδελφο να θέλει το λόγο. Και ο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κόνη. Καλημέρα σας. Μας με κόνια. Και έχουμε σε αυτό το θέμα του, του, του καινούριου ταμείου στη Γενική Διεύθυνση για την Αλληλεία, το Ταμείο για τα Θεσσαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλληλεία. Δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο καινούργιο να πούμε, απλώς να ξεκαθαρίσουμε το ότι η πρόταση αυτή τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να βοηθηθούν οι κοινότητες των Αλληλείων και έχουμε και ένα κεφάλαιο το οποίο α, ακριβώς αφορά αυτό το θέμα σε σχέση με τη φάση αυτή στην οποία τώρα βρισκόμαστε στο σχέδιο ε, κειμένου και στις ε, διαπραγματεύσεις έχουμε θίξει το ζήτημα της ε, αηφόρου ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και τονίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο το πόσο σημαντικά είναι αυτά. Επίσης λέμε ότι με αυτό το ταμείο έχουμε ε, μια σειρά από ενδυνάμει εφικτά μέτρα και με συνδιαχείριση είπαμε ότι θα πρέπει να αποφασιστεί ποια μέτρα θα υιοθετηθούν και ποια όχι. Ελπίζουμε επομένω ότι τα κρατη θα αποφασίσουν ανάλογα και στα πλαίσια ε, της, του ρόλου μας και της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελπίζουμε κάθε τον τρόπο να συνεχίσουμε να προβάλλουμε αυτές τις προτεραιότητες. Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Και νομίζουμε ότι τώρα βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, σε μια κρίσιμη εξέλιξη σε σχέση με το προηγούμενο πρωτοδοτικό μέσο, γιατί καταργήθηκαν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ αδόκιμα αυτά που αφορούν τον στόλο. Τη αποσύρση των ελευτικών αντικαταστάσεων κινητήρων κλπ. Ε, γι' αυτό και θεωρούμε ότι ε, με το που σταμάτησαν αυτές οι άμεσες επιδοτήσεις, τα κράτη-μέλη πρόκειται να εστιάσουν την προσοχή τους στην αηφόρα ανάπτυξη στις ε, αλήθικες περιοχές. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ όλους τους έλεγαν τον λόγο. Θα λάβω υπόψη όλα αυτά τα οποία είπαν. Πολύ σημαντικό να έχουμε τροπολογίες, κυρίως όσον αφορά τους νέους. Νομίζω ότι με τους ε, σκιώδες πρόκειται να εργαστούμε καλά, να συνεργαστούμε και να έχουμε σε κατάληξη. Ευχαριστούμε πολύ. Τροπολογίε. 10 Ιουλίου το μεσημέρι, 18 Ιουλίου θα συζητήσουμε και του συνδεσμούς 8 και 9 και θα ψηφιστούν στην ε, Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Επιτροπή Αλίας, 28 Νοεμβρίου θα εγκρίνει το θέμα και, και θα πάει μετά η έκθεση εκείνη στην ορμένα του Ιανουαρίου. Σήμερα το καινούργιο πλαίσιο, κάθε επιτροπή έχει άλλους ρυθμούς τώρα. Παρακαλώ όλες τις πολιτικές ομάδες να κινητοποιήσουν τα μέλη τους, να στείλουν ένα ένα mail για την 11.30 ώρα. Θα έρθει εδώ ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Οργανώσης Εργασίας. Να είναι γεμάτη η αίθουσα, όσο γίνεται περισσότερα ε, μέλη της Επιτροπής. Γιατί είναι σημαντικό. Λόγω των σχέσεων που θέλουμε να έχουμε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας. Ε, επειδή είναι σημείο αναφοράς για μας. Κλείσαμε επομένω τη συζήτηση του σημείου παριθμού 18 της μέσης διατάξεως και πάμε τώρα στο 19. Και έχουμε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιασλοβιέτσκα. Θα μας παρουσιάσει στα πλαίσια αυτής της έκθεσης ε, ίδιας πρωτοβουλίας το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως απάντηση στην κρίση. Να μας πει δύο λόγια τις 154 τροπολογίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τις 154 τροπολογίες τις οποίες έχετε υποβάλει για το έγγραφό μου. Ήσασταν πάρα πολύ δραστήριοι και αυτό αποδεικτεί πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Πράγμα το οποίο ίσως δεν αντικατοπτρίζεται στις παρουσίες ε, εδώ αλλά στον αριθμό των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Ε, νομίζω ότι το πιο βασικό θέμα εδώ είναι η εφαρμογή. Οπότε όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής πρέπει να εμπλακούν στο τι θα αποφασιστεί σχετικά με το έγγραφο αυτό και γι' αυτό θέλω το κείμενό μου να αντικατοπτρίζει τις περισσότερες ε, θετικές ιδέες που παρουσίασαν οι συνάδελφοι. Θέλω να παρουσιάσω ορισμένα σχόλια και να σας πω ότι η πλειοψηφία θα, ε, ε, των τροπολογιών θα υιοθετηθούν αλλά σχετικά με τις διαγραφές για το την τροπολογία 145 ή αυτοί οι οποίοι απορρίπτουν την αιτιολογία η οποία προβλέπεται στην τροπολογία 14 και 15 όσον αφορά την ε, κοινωνική ε, φτώχεια. Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το επηρεάσουμε δια δράσεων στην αγορά εργασίας παραδοσιακές. Ε, ε, δεν φτάνει δηλαδή η ενίσχυση το, της, παρασυ, παραδοσιακής βοηθείας στην ε, ε, αγορά εργασίας. Θα πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και όλα τα θέματα που μιλούν για σταθερότητα, για περισσότερη δραστηριοποίηση των πολιτών που θα πρέπει να ψάξουν ενεργά για δουλειές, ε, όλα τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βρίσκουν απολύτως σύμφωνοι. Πιστεύω όμως ότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο όπου η παραδοσιακή μορφή του κράτους προνοίας δεν επαρκεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενεργό κράτος προνοίας και να μιλήσουμε για τα στοιχεία που ε, επιτρέπουν να αλλάξει η κατάσταση στην αγορά εργασίας και συμφωνώ με τις ε, απόψεις των συναδέλφων επί του θέματος αυτού. Ε, σχετικά με τις τροπολογίες που θα περιλάβω ή στις τροπολογίες 7, 8, 9, 10 και 11 ε, σχετικά με την τροπολογία 11 δεν είμαι βέβαιη ότι υπάρχει μία κρίση ανταγωνισμού ε, για τις 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28 και 30 31, 33, 34 και 35 και τονίζω εδώ την 33 γιατί δεν ξέρω εάν πρέπει να επενδύσουμε μόνο στην παιδεία και ότι αυτό, αυτή είναι η πανάκια για όλα τα δεινά της αγοράς εργασίας αλλά νομίζω ότι αυτή η τροπολογία πρέπει να περιληφθεί στη συμβιβαστική, στο συμβιβαστικό κείμενο. 37-39 επίσης θα συμπεριληφθούν. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την μαύρη αγορά της εργασίας, την παράνομη εργασία και ευχαριστώ τον κύριο Πουπάκη που μου τόνισε αυτό το σημείο, δηλαδή ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις παράνομες μορφές εργασίας. Κατά τα άλλα είμαι ικανοποιημένος διότι ο συνάδελφος που είναι συντάκτης τονίζει την σημασία των, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα πρέπει και αυτές να συμπεριληφθούν στις διεργασίες ε, σχετικά με το 53 ε, έως 57-58 θα περιληφθούν επίσης στο συμβιβασμό στην τροπολογία 60 η κυρία Σάια ε, προτείνει να συνδράμουμε τα κράτη που είναι σε κρίσιμη θέση σχετικά με το κοινωνικό σύμφωνο απασχόλησης αλλά δεν νομίζω ότι το να είναι κανείς σε κρίσιμη κατάσταση επαρκεί σαν κριτήριο ε, τροπολογίες από 60 έως 70. Επίσης συμφωνώ για το 72 θέλω κάποια διευκρίνηση διότι λέγεται ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ικανοποιητικό εισόδημα για όσους ε, ε, το έχουν ανάγκη. Ε, το 77 ε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για βιώσιμες νέες θέσεις εργασίας διότι υπάρχουν και πολλές ασταθείς θέσεις εργασίας τώρα που θα έπρεπε να περιληφθούν στο μέτρο αυτό. Ε, ε, ε, οι τροπολογίες 80 ε, μέχρι 100. Στο 91 θα ήθελα μία διευκρίνηση διότι δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείται όταν μιλάτε για επαγωγικές συνθήκες. Conducive conditions. Ε, το 93 είναι ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερος και πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις 99 προληπτικά μέτρα που προτείνονται τα δέχομαι 101 έως 106 έως και 111 107. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε τον όρο με απασχόληση και να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι να επιτύχουμε αντί τι θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Αν δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας βεβαίως η ανεργία θα μειωθεί και αυτό είναι πιο θετικό. Όσον αφορά το 113 θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπάχαν μπορεί να μου διευκρινίσει τι εννοεί ε, για απασχόληση ε, για ε, ανεκπαίδευτους ή ανεπαρκώς εκπαιδευμένους εργαζομένους. Σχετικά με τις τροπολογίες της κυρίας Γκιόνς θα ήθελα να μου πει τι εννοεί όταν μιλά να δημιουργηθεί η σωστή ε, ατμόσφαιρα στα σχολεία. Δηλαδή θα μπορούν έτσι οι νέοι να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας 123 και 124. Ε, με βρίσκουν σύμφωνοι αλλά στο 124 βλέπω ότι οι κοινωνικές επενδύσεις θα πρέπει να προσπαθήσουν να ε, περιλάβουν ε, και την περίθαλψη των ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικά ιδρύματα. Δεν το καταλαβαίνω περαιτέρω 134 θέλω να ζητήσω μία διευκρίνηση γιατί βλέπω ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να ενθαρρυνθούν να εργαστούν με τα κατάλληλα μέσα. Τι εννοείται όταν μιλάμε για κατάλληλα μέσα. 100 40 έως 146 επίσης με βρίσκουν σύμφωνοι. 146 και 149 είναι τροπολογίες οι οποίες με ικανοποιούν διότι επεκτείνουν αυτά που είχαν προταθεί στο αρχικό κείμενο και ε, ο συντάκτης αναφέρεται εις ε, την συμμετοχή στα μέτρα και στο σύμφωνο επενδύσεων. Δεν ξέρω βέβαια ε, πώς εσείς διαβλέπετε τις πηγές για κοινωνικές επενδύσεις. Ευχαριστώ όλους για τις τροπολογίες, συμπληρώσατε τη δουλειά μου και επειδή πρόκειται απλώς για μία γνωμοδότηση δεν μπόρεσα στο αρχικό μου κείμενο να περιλάβω όλες αυτές τις ιδέες αλλά αυτή την εβδομάδα θα επεξεργαστώ τις συμβιβαστικές τροπολογίες θα τις στείλω στους κοιόδης και σε όλους τους ενδιαφερομένους συναδέλφους κατά τρόπον ώστε να μπορέσετε να προωθήσετε τις θέσεις μου στα κράτη-μέλη. Κυρία Παπαδοπούλου, αλλά πριν δώσω το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου, να υποδεχτώ εδώ στο βάθος της αίθουσας μία αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου της ε, Gironde, της, Ακικτά, ε, που ήρθαν εδώ στο Κοινοβούλιο για να δούνε πώς εργαζόμαστε, πώς χρησιμοποιούμε το FSE και σας ευχαριστούμε που θα μείνετε μαζί μας μέχρι για τα επόμενα 20 λεπτά που θα έρθει και ο νέος πρόεδρος διευθυντής της ΔΟΕ, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να συγχαρώ την εισηγήτρια εν ονόματι των σοσιαλιστών και να εκφράσω την εκτίμησή μου διότι ορισμένα από τα μέλη του ΕΚΤ όπως και η εισηγήτρια που προέρχεται από την Πολωνία αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια δεν μπορεί μόνη της να επιλύσει την οικονομική κρίση. Ε, προ λίγων λεπτών άκουσα και ε, σχεδόν ε, οι μισές από τις τροπολογίες των σοσιαλιστών επί συνόλου 28 θα περιληφθούν στις συμβασικές τροπολογίες και πιστεύουμε ότι εάν υιοθετηθούν όντως θα συμπληρώσουν αυτή την έκθεση. Ε, στις τροπολογίες μας λέμε ότι η οικονομική κρίση όντως έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ε, και στις οικονομίες αλλά και στις δημόσιες και κοινωνικές επενδύσεις στην Ευρώπη και τονίζουμε στην τροπολογία 13 και λέμε ότι τα κρατικά μέτρα τα οποία επεδίνωσαν την κατάσταση στην Ευρώπη δεν επαρκούν, θα πρέπει να υπερβούν την ε, ε, κοινωνική πειθαρχία ε, και τη δημοσιονομική πειθαρχία και θα χρειαστεί ε, η βελτίωση του προϋπολογισμού να συνδυαστεί με μέτρα επενδυτικά, αναπτυξιακά και βελτίωση της απασχόλησης συγχρόνως με μεγαλύτερη προσήλωση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους της στρατηγικής για το 2020 διότι η κοινωνική απασχόληση στην ατζέντα του 2020 δεν έχει εφαρμοστεί από τα περισσότερα κράτη-μέλη και επιπλέον η ανεργία αυξήθηκε 7,1% το 2008 σε 12% το 2012 και βλέπουμε ότι 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κινδυνεύουν με φτώχεια και ανεργία των νέων. Όλα αυτά τα θέματα θίγονται στις τροπολογίες μας και υπάρχουν πάρα πολλοί ε, νέοι οι οποίοι ζουν σε ανεργανικά νοικακυριά και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει ικανοποιητική προσφορά εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλα αυτά, πιστεύω ότι οι επεμβάσεις στο κράτος προνοίας δεν έχουν επιλύσει το θέμα της κρίσεως, οδήγησαν σε μία μείωση των εισοδημάτων και χρειάζονται πάρα πολλά μέτρα πέραν της λιτότητος για να προβληθούν οι δεξιότητες ε, της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένες εστιασμένες κοινωνικές ε, επενδύσεις στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 για να δημιουργηθούν θέσεις υψηλού επίπεδου και ποιοτικέ ε, ε, στα πλαίσια αυτά και με ικανοποιητικά μισθός και με βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε συνεργασία με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να προωθήσουμε την ισορροπία μεταξύ ασφαλείας και ευελιξίας στην αγορά εργασίας μειώνοντας την ε, εξάρτηση ε, από κοινωνικούς πόρους. Αυτό είναι ε, το, η πεμπτουσία των 28 τροπολογιών που υπέβαλε η πολιτική μου ομάδα και την άλλη εβδομάδα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διαβολευτούμε ε, τους υπόλοιπους εισηγητές των πολιτικών ομάδων για να τονίσουμε ορισμένες πτυχές στην έκθεση η οποία καταρτίστηκε. Η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Είμαι η σκιώδη εισηγήτρια. Μάλλον η σκιώδη συγγνώμη δεν είναι εδώ, αλλά θα της πω τι είπε Εισηγητρία, και γιατί έχουμε εδώ πέρα μια σειρά από τροπολογίε και ακριβώ ε, και αυτό που είπατε και εσεί να υπάρχει κάποιο είδου ε, θετική διατύπωση όσον αφορά ε, την, την ανεργία των νέων και σας ευχαριστούμε πάντως για τη θετική σας απόκριση για το 146. Ζητείτε εδώ να διευκρινίσουμε κάποια σημεία και σε άλλες τροπολογίες. 72 όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια. Θα, θα, ζητήσω από την ε, συνάδελφο να σας τα διευκρινίσει και επίσης όσον αφορά την τέταρτη παράγραφο και εμείς το ξαναείδαμε και ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς όσον αφορά κάποια στοιχεία που θα πρέπει να αφορούν αυτήν, αυτήν την ε, θετική κινητοποίηση. Πάντως συμφωνούμε με τη δική σας γραμμή και περιμένουμε πώς και πώς να συνεργαστούμε για τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που παρουσίασαν. Σας ευχαριστώ για τις ε, προτάσεις. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο η πολωνική αντιπροσωπεία του ΕΛΚ. Όλο το ΕΛΚ, όλη η χριστιανοδημοκρατική οικογένεια πιστεύει ότι η εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής είναι πολύ σημαντική. Εμείς θέλουμε κυρίως να αλλάξουμε την οτροπία μας. Εγώ αναφέρομαι σε αυτό στην έκθεσή μου Θέλουμε το κοινωνικό στα κράτος να είναι ένα κράτος το οποίο ε, προσδίδει, ενδυναμώνει την ε, κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο πλούσια, δεν μπορεί να επενδύει μόνο σε αυτούς τους πολίτες ε, που ζουν στη φτώχεια. Εμείς πρέπει να παρέμβουμε όπως κάνουν και, τα κράτη, και οι Ηνωμένε Πολιτείες Πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι και πρέπει να αισθάνονται ευθύνοι και έναντι των παιδιών τους και έναντι των γονιών τους. Και για να μπορέσουν να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες πρέπει να είναι ενεργοί. Εμείς θα θέλαμε η κοινωνία μας να είναι μια δυναμική, μια ενεργός κοινωνία, διότι έχουμε άτομα με μεγάλες δυνατότητες, οι νέοι κυρίως που μπορούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να βρουν μια θέση στις Ηνωμένε Πολιτείες ή στην Κίνα. Ε, λυπούμε βέβαια για αυτήν τη μετανάστευση, για αυτήν τη μοίρα. Θα θέλαμε οι νέοι μας να είναι πιο δυναμικοί δεν θα θέλαμε να υποστηρίξουμε μόνο αυτούς οι οποίοι ζουν σε μια κατάσταση παινίας, αλλά θέλουμε να δώσουμε δυναμική, να ενεργοποιήσουμε τα άτομα στα διάφορα κράτη-μέλη. Η κοινωνική πολιτική οδηγεί πολλές φορές σε μια αύξηση της στόχιας και όχι στο αντίθετο. Χαίρομαι λοιπόν που αυτή η έκθεση έγινε δεκτή με μεγάλη υποστήριξη. Θα μπορούσα, πιστεύω ότι είναι δυνατόν να ετοιμάσουμε από κοινού ένα καλό έγγραφο που θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε αυτή την οτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουμε σε αυτές τις κοινωνικές επενδύσεις. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες το 10 και θα τις ψηφίσουμε. Λοιπόν, διακόπτω τώρα τη συνεδρίαση μέχρι τις 11.30 που θα και αυτό θα, περιμένοντάς σας να ξανάρθετε μετά για να ακούσετε τον νέο Γενικό Διευθυντή της ε, ΔΟΕ, τον κύριο Ρίντερ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και μεγάλη μου τιμή που υποδέχομαι τον Γκί Ράιντερ, τον ε, φρέσκο τον νεοεκλεγμένο Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ 28 Μαΐου ε, εκλεγήκατε. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να είμαστε από τους πρώτους που έρχεστε να συναντήσετε. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε αυτές τις ανταλλαγές για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα θέλω εξ ονόματος όλης της Επιτροπής να σας ε, καλωσορίσω, το έκανα γραπτός, ε, το ξαναλέω και προφορικά. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός, ήταν πολύ σημαντικός ο αριθμός ε, των υποψηφίων και ο γύρος ψηφοφοριών επίσης ε, πολλές φορές, πολλαπλώς. Η... Όλη σας η ιστορία η προσωπική σας ιστορία και η εμπειρία σας επέτρεψαν να κερδίσετε. Σας εύχομαι για την άσκηση αυτής της τόσο ωραίας εντολής, αυτήν την τόσο δύσκολη στιγμή, ό,τι καλύτερο. Οι σχέσεις που έχουμε η Επιτροπή μας με την οργάνωσή σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς ε, θέλουμε να, να τονίσουμε τις ε, σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και ΔΟΕ. οι βασικές συμφωνίες δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε σε μία ιστορική στιγμή και οι αξίες των οποίων φορέας είναι η ΔΟΕ είναι αξίες που όλοι τις συμμεριζόμαστε δεν λαμβάνονται όμως υπόψη από όλα τα κράτη-μέλη. Διότι λένε ότι ορίστε αυτό είναι για τις αναδυόμενες χώρες, για τις ε, υπανάπτυξη χώρες και εμείς είμαστε υπεράνω όλων. Εμεί θεωρούμε ότι οι Ευρωπαίοι όχι απλώς δεν, είναι υπεράνω, δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου, αλλά πρέπει να, δείχνουν και το, να δίνουν και το καλό παράδειγμα. Και θέλουμε όλες οι βασικές συμφωνίες να εφαρμόζονται από όλου και να τις επικυρώσουμε. Επίσης, μέσα στο πλαίσιο της κρίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχετε στην όλη συζήτηση για την παγκόσμια διακυβέρνηση, για το ρόλο της ΠΟΕ αλλά και η ανάλυση και πραγματογνωμοσύνη για το κοινωνικό σοκ το οποίο δημιουργεί η κοινωνικό χρηματοπιστωτική κρίση. Και η συνεργασία σας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καρποφόρα κατά τη γνώμη μας. Εμείς θεωρούμε ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλάβαμε την πρωτοβουλία, θα θυμάστε πριν από τη Γενική σας Συνέλευση, να έρθουμε να ε, ενισχύσουμε τις εργασίες της και πιο συγκεκριμένα τη Σύμβαση για την Οικιακή Εργασία. Και θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει μία συνέργεια την οποία θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε και να την αναπτύξουμε. Πριν σας δώσω το λόγο θέλω να χαιρετήσω επίσης και τον προκάτοχό σας, χάρη του οποίου ξεκινήσαμε όλη αυτή την εξαιρετική συνεργασία, την οποία ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε και θα αναπτύξουμε με θυμόν. Η, εργα... η αντιπροσωπεία μας ε, έχει αρχίσει και ευχαριστιέται με αυτές τις ε, μετακινήσεις στη, Γενά, στη Γενέβη, οπότε τώρα σας στέλνουμε το ασανσέρ για να αρχίσετε να μετακινήσετε και εσείς προς τις Βρυξέλλες. Σας δίνω το λόγο για την εισαγωγή σας. Και μετά θα ξεκινήσουν οι ερωταπαντήσεις με τους βουλευτές. Καλημέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για αυτή την εισαγωγή και κυρίως σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα το πρωί. Και θα ήθελα να σας πω για να ξεκινήσω, αλλά δεν ξεκινάω. Στην ουσία συνεχίζω τον διάλογο μεταξύ του, της Διεθνούς Οργάνωσης Υγείας ε, και εσάς και να προβληματιστούμε από κοινού, γιατί νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση του να συσκεπτόμεθα για το τι θα γίνει αυτός ο διάλογος, πώς θα προωθηθεί μέσα σε αυτές τις περιστάσεις, οι οποίες, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πάρα πολύ δύσκολες για, για την αγορά της απασχόλησης, πολύ προβληματικές, είναι κάποιες ε, συνθήκες τις οποίες ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε την συνεργασία μεταξύ της ΔΟΕ και της Επιτροπής σας. Για να σου πω βλέπει η Γενέβη τα πράγματα που αναφέρατε. Πρώτα πρώτα, σας αναφέρω ότι η ΔΟΕ εκτιμά πάρα πολύ την συνεχή και συνεπή υποστήριξη εκ μέρου σας όσον αφορά να υπάρχει μια ατζέντα ουσιαστική για την απασχόληση και να γίνεται αυτή η ατζέντα ε, δράση και πράξη στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Δεν είναι προκάτοχο, είναι ο γενικό διευθυντή που είχε μιλήσει στο Κοινοβούλιο, νομίζω είχε μιλήσει ε, τον ε, Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, γιατί είναι νομίζω φυσική ούτως πίν. Έρχεται φυσικά η συνεργασία μας, έχουμε κοινέ αξίε κοινού στόχους και σκοπούς, οπότε είναι φυσικό να συνεργαστούμε για την υλοποίησή τους. Τώρα, θα ήθελα να σας θέσω ορισμένα ζητήματα και να σας πω κάποιες προτάσεις που θα πρέπει να από κοινού να μας απασχολήσουν. Έχουμε ιστορία 90 ετών. Η ΔΟΕ ανέκαθεν ήταν σε θέση να υπολογίζει στη βοήθεια των Ευρωπαίων να είναι οι ατμομηχανές, οι πρωτοπόροι. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι θέλουμε την τριμερή συνεργασία, τον κοινωνικό διάλογο και αυτό το πνεύμα που μας διαπνέει εκφράζεται με το ότι η οικονομική ανάπτυξη φέρνει κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο. Αυτό είναι η ουσία του πνεύματος μας διαπνέει και επί 90 έτη θα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι για να είμαστε ειλικρινεί, όσο και να είναι πολύπλοκα τα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη, η Ευρώπη είναι κατεξοχήν το μέρος όπου υλοποιούμε αυτούς μας τους στόχους. Εκεί έχουμε πετύχει ιστορικά σε εξαιρετικό βαθμό ε, αυτά τα οποία θέλουν την κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο. Σήμερα δε, νομίζω δε, ότι είναι κάτι το μοναδικό στην ιστορία μας. Έχουμε κάτι σαν αντιστροφή της, της συνήθους τάξης των πραγμάτων. Βλέπουμε, διαπιστώνουμε. Να μαστίζεται η Ευρώπη από κρίση. Είναι το επίκεντρο της παγκόσμιας κρίσης. Και όποιος παρατήρησε τι έγινε στο Λοσκάβος στην, στο, στην G20 τότε καταλαβαίνετε τι είπε είναι πολύ σοβαρή στην Ευρώπη και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις να και το παράδοξο κάποιες χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν εμπνευστεί από την Ευρώπη ενώ για τις αναδυόμενες χώρες πολλές λοιπόν στον αναπτυσσόμενο κόσμο σήμερα έχουν ευκαιρίες γιατί συνεχίζεται ο δυναμισμός τους και γι' αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πετύχουν μια κοινωνική δικαιοσύνη, μια κοινωνική πρόοδο που δεν την είχαν στο παρελθόν. Οπότε γι' αυτό το λόγο και τώρα μπορεί να δει κανεί τι γίνεται στη Λατινική Αμερική, όπου υπάρχουν παράλληλα και άλλοι και εκεί ευκαιρίε, ώστε να προχωρήσουν για κοινωνική πρόοδο. Και αυτό δεν είναι μόνο οι δυνατότητε. Οι δυνατότητε να υλοποιηθούν. Και σε σχέση με την Ασία έχουμε πάντα κάποιες ε, αμφιβολίες και πολλές φορές δεν έχουμε δώσει την προσοχή που χρειάζεται και εκεί πέρα. Δεν έχουμε μόνο ευκαιρίες, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη τάση σε αυτές τις χώρες και σε αυτές τις χώρες να εντάξουν τώρα και την Ινδία. Να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κάποιες κοινωνικές, πολιτικές και τα ελλείμματά τους. Τώρα είναι στοιχείο της κρατικής πολιτικής η Κίνα να δίνει περισσότερα στους εργαζομένους. Και έχουν βάσιμους λόγους. Έχει να κάνει με τις ανισορροπίες της δικής τους οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας. Βλέπετε όμως τώρα εδώ ότι υπάρχει αυτή η ατζέντα κατά την οποία ε, δίνεται άλλη θέση. Καλύτερο τρομερίδιο στην ευημερία προς τους εργαζόμενους. Να, επομένω, πώ σιγά σιγά φτιάχνουν και ένα σύστημα αποτελεσματική κοινωνική πρόνοια για πρώτη φορά. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανεί. Και δεν σα ε, εκπλήσω το ίδιο το ίδιο και στην Αφρική. Τα ξέρετε. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαν μπει στη φάση τη αγρονάπτυξη. Τώρα όμω και εκείνοι κινούνται προ την κοινωνική πρόοδο. Και επομένω, κατά κάποιο τρόπο ακολουθούν το μονοπάτι που χάραξε η Ευρώπη. Εδώ και καιρό. Ταυτόχρονα η Ευρώπη ε, βρίσκεται στον αντίποδο, όπου οι κοινωνικές κατακτήσεις πολλών δεκαετιών, κοινωνική πρόοδος που πετύχανε κάποιοι σαν και σε χώρους όπως εδώ, τώρα αμφισβητούνται. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο να διατηρηθούν. Βλέπετε επομένως πώς έχετε τον κόσμο αυτή της απασχόλησης, αυτές τις συζητήσεις, με τρόπο που δεν μας είναι τόσο οικείος. Άρα, τι να συμπεράνουμε από αυτά, αυτή την πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει παντού σκοτάδι και απεσιοδοξία. Δεύτερο. ό,τι και να γίνει επόμενη δεκαετία, η Ευρώπη θα είναι ο πρωταγωνιστής. Μην έχετε αμφιβολίες. Βέβαια, εσείς τώρα φέρετε το βάρος αυτού του καινούργιου ρόλου. Η ΔΟΕ τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπατε διάφορα πρόεδρε. Είπατε για τις αξίες, τα θέματα των θέματα των δικαιωμάτων και έχετε δίκιο 100%. Η συγκρότηση του, της ΔΟΕ ταυτίζεται με την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε οκτώ τέτοιες ε, συμβάσεις, συμφωνίες, συνθήκες και οι επιδόσεις της Ευρώπης είναι πάρα πολύ αξιόλογες της Πίζας, η μία ακόμα, μη κυρωθήσα σύμβαση, τέλος πάντων. Καλείστε να εφαρμόσετε ό,τι πρέπει, ε, θέμα το οποίο είναι πολύ συζητήσιμο, αλλά πάντως η ΔΟΕ με το σύστημα που ισχύει τώρα και δικαιολογημένα είναι σε θέση να αναλάβει δράση. Και Τώρα πρόσφατα η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση απέδωσε καρπούς. Και μιλώ για την Μπούρμα, την Μιανουάρ. Δράσαμε, επιμείναμε για 15 χρόνια να κάνουμε κάτι αυτή την ε, χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρπαξε την ευκαιρία και όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο. Οπότε σήμερα αυτή η χώρα μπορεί να έχει δεκαλιστικούς εργαζομένων κλπ. Είναι έτοιμη να μπει ξανά στην ε, διεθνή κοινότητα να κάνει τον δημοκρατικό μετασχηματισμό. Φοβερή, φοβερό επίτευγμα. Κατά πολύ αυτό οφείλεται στη δράση του της ΔΟΕ και στο πόσο πρόθυμη ήταν η Ευρώπη να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να φέρει την αλλαγή. Αυτό το λέω που και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ανταπόκριση τώρα για την κρίση, για τις κρίσεις και εδώ ε, πάρα πολύ καλά τα πήγαμε στη συνεργασία μας το 2009 όπως τα γνωρίζετε η ΔΟΕ υιοθέτησε αυτό το τριμερές ε, έγγραφο, τριμερή συμφωνία όπου είπαμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιδράσουν στην κρίση το 2009. Τότε που οι απαρχές της κρίσης σιγά σιγά γίνοντουσαν σαφείς και καταλαβαίναμε ότι πρόκειται για κοινωνική παγκόσμια κρίση, οικονομία, απασχόληση, άρχισαν να υφίστανται τις συνέπειες. Και θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία, το Global Jobs Pact όπως ονομάζεται, θα είναι ένα λιθαράκι παραπάνω στις προσπαθίες μας η απασχόληση, δημιουργία θέσεων εργασία, είναι στο επίκεντρο της απόκρισής μας στην κρίση, της αντίδρασής μας. Κανένας δεν πρέπει να θεωρεί ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει την κρίση αν δεν έχει κοινωνικό διάλογο και αν παραβιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτά τα θέματα παραμένουν καυτά και βλέπουμε ε, τα σκαμπανεβάσματα από το 2008. Τον Εύρω 2008, τότε, τότε ο Τζορτζ Μπούς, ο νεότερος, συγκρότησε την ομάδα των G20. Άρα θα πρέπει να κάνουμε, λέγαμε, μέχρι το 2008 να, να, να κάνουμε μικρές αλλαγές στο χρηματοπιστικό σύστημα μέχρι το 2009 πάλι στο Λονδίνο τον, τον, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, Λονδίνο, Πίτσμπεργκ, οι G20 τα είπαν αυτά και μέχρι τον Οκτώβριο 2009, λίγο μετά το Global Jobs Pact το δικό μας, ήταν σαφές του g ότι η απασχόληση ήταν στο επίκεντρο της ανάκαμψη. Κατόπιν ήρθε η κρίση του χρέους στην Ευρώπη και έτσι ξαναπήγαμε στη μελέτη των δημοσιονομικών στο Μεξικό. Τώρα βλέπουμε ότι ο τροχός ξαναγύρισε προς τα θέματα απασχόλησης. Και φυσικά πάλι είχαμε και αλλαγή στο τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο τοπίο. Πέρασαν 34 χρόνια επομένω και αυτά τα σκαμπανεβάσματα, χρηματοοικονομικά, απασχόληση, όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν ε, αξιοπιστία, ε, δόκιμη πολιτική, σωστή, γερή, δυναμική, αντίδραση στην κρίση και επομένως μαζί θα πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε μεγαλύτερη συνέπεια, πώς θα γίνουμε ικανότεροι να δούμε όλες τις, τις πλευρές της κρίσης, όλες τις διαστάσεις που θα πρέπει να έχει και η αντίδραση στην κρίση. Φυσικά και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο κανείς να ε, κάνει συνέχεια αυτές τις συζητήσεις για τη λιτότητα κλπ. Πρέπει όμως να αναζητήσουμε το σωστό μείγμα πολιτικής, να έχουμε εξυγίανση δημοσιονομική, αλλά να έχουμε και θέσεις εργασίας. Και ταυτόχρονα να κάνουμε και την κοινωνική μας πολιτική. Να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις που είδαμε ότι έχουν τέτοιες διαστάσεις που δεν περιμένουμε τίποτα. Να, ποιες είναι οι προκλήσεις. Δεν μπορούμε να τις παρεβλέψουμε. Θα πρέπει. Επομένως, προς τα εκεί να κατατείνουν οι προσπάθειές μας. Και το μήνυμα ποιο είναι για σήμερα, Πρόεδρε. Η ΔΟΕ ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ να συνεργαστεί με εσά, με την Επιτροπή σας, με την Ένωση. Και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αναφέρατε και το δυνατό το 2010. Όντως είχαμε θετική συνεργασία, έγινε η πρώτη συνάντηση ιστορικής σημασία για κρυβάσουμε τους παράλληλους και όχι άλλους συγκρουόμενους στόχους. Χρηματοπιστωτική τάξη και καλύτερη απασχόληση. Νομίζω ότι κάναμε βήματα πρόοδο. άλλο που συνδέεται με το προηγούμενο. Ελπίζω ότι η επίδραση της ΔΟΕ και η συμβολή μας στο έργο σας να θεωρείται σημαντικό. Νομίζω ότι προκύπτει αυτό. Και αυτό το οποίο θέλουν τα τρία μέρη, τρεις πλευρές, τρεις παράγοντες, στη ΔΟΕ είναι ότι αυτά όλα θα πρέπει να την υπόψη για την κοινωνική πολιτική, μια που η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι ο ρόλο που έχουμε διαδραματίσει, όποιο να ήταν αυτό, είναι ότι ήμασταν ο πυροσβέστης όταν έπιανε φωτιά. Πήγα στην Ελλάδα. Πήγα και ξαναπήγα στα πλαίσια των, των, των πακέτων τη Τρόικα. Μα φωνάξανε για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε των πολιτικών που αποφασιζόντουσαν αλλού. Εμεί δεν είχαμε ρόλο στι πολιτικέ, δεν είχαμε γνώμη. Μα φωνάξαν όμω για να σβήσουμε την κοινωνική πυρκαγιά που άναψαν αυτά τα μέτρα. Και αυτό το οποίο θέλω να σα πω είναι ότι πρέπει να το διερευνήσουμε. Και αύριο θα πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια που θα είχα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και απαιτείται να ενεργήσουμε άμεσα. Όμως, υπάρχει κάτι το οποίο θα το σημειώσετε στην ατζέντα τον Απρίλιο του χρόνου. Θα πάμε στην περιφερειακή συνάντηση, αυτό την τετραετή συνάντηση αυτή, στο Όσλο. Μας καλεί η κυβέρνηση της Νορβηγίας. Πρόκειται για μια εκδήλωση βασική, κλασική. Όμως τώρα τα πράγματα πιέζουν και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δράσουμε, να συνεργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ε, διάσκεψη για να μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποια από τα εκκρεμούντα θέματα, τις προκλήσεις. Να μην υποτιμήσουμε αυτά που πετύχαμε στο παρελθόν. Εμείς πάντα έχουμε πάντως το καθήκον να κάνουμε καλύτερα από όσα κάνανε οι παλιότεροι. Όλα αυτά επομένω θα ωφελήσουν το μέλλον τη δράση της ΕΔΟΕ και εσά και αυτού που εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δώσατε να σα πω αυτά τα λόγια. Ε, ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η ανταλλαγή απόψεων και σήμερα αλλά και στο μέλλον. Ε, ευχαριστώ για όλα όσα αναφέρατε για το ρόλο της οργάνωσής σας Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω της Τρόικας. Ξέρετε ότι σε αυτό το κοινοβούλιο ψηφίσαμε ήδη την ιδέα ότι θα έπρεπε να συμμετέχετε στις διάφορες Τρόικες. Αυτό το είχαμε ψηφίσει σε μία έκθεση της οποίας ήμουν συντάκτης και τότε είχαμε πει ότι θα έπρεπε να συμμετέχετε στις διάφορες Τρόικα. ο κύριος ορί. και μετά ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα, θα ήθελα να χαιρετήσω τον Γενικό Διευθυντή, όχι ως απλά και μόνο ως νεοκλεγμένο διευθυντή αλλά και ως συνεργάτης του κυρίου Σωμαβίγια ε, μπόρεσε να παρακολουθήσει από κοντά τις εργασίες μας. Έχουμε ε, πλεονεκτικές ε, σχέσεις μαζί του. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Εξ ονόματος του ΕΛΚ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω που εκλεγήκατε Γενικός Διευθυντής. Βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, είμαστε συνομιλητές εκφύσεως. η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και όλα τα επίσημα έγγραφα του Κοινοβουλίου εξάρουν τον ρόλο της ΔΟΕ. Αυτά τα οποία μας αναφέρατε αποδεικνύουν ότι εσείς έχετε στη ΔΟΕ μια ευρύτερη εικόνα, μια ευρύτερο βλέμμα ε, για την Αφρική, για την Κίνα, για όλες τις περιοχές του κόσμου. πολύ πιο αντικειμενική ματιά από αυτή την οποία έχουμε εμείς έναντι των ενδυνάμει ανταγωνιστών μας και αυτή σας η αντικειμενικότητα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Η συνεργασία σας ε, είναι πολύ σημαντική. Ε, πριν από μερικές δεκαετίες η ΔΟΕ ασχολιόταν με το θέμα της Βυρμανίας. Αληθεύει ότι ζούμε κρίση στον κόσμο πρώτη προτεραιότητα για μας είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση και πρέπει να έχουμε ένα βλέμμα πολύ πιο κοινωνικά ευαισθητοποιημένο. Η κοινωνική κατάσταση σήμερα οδηγεί σε μία αλλαγή του πνεύματος του κοινού. Και ο τομέας αυτός είναι ένας τομέας όπου οι μηχανισμοί που ισχύουν εδώ και 90 χρόνια στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας μας ενθαρρύνουν για να είμαστε υπομονεκτικοί και ανεκτικοί και πιστεύουμε ότι μία συνεργασία στην καταπολέμηση της κρίσης θα μπορέσει να μας ε, είναι πολύ χρήσιμη. Επιπλέον υπάρχει κι άλλος ένας τομέας που πρέπει να μας ε, απασχολήσει είναι η συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πρέπει να θεωρήσουμε ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και βλέπουμε ότι παρόλη τη βοήθεια που χορήγησε ε, το Ταμείο αυτό ούτε αύξησε τη δημοτικότητά του αλλά αντιθέτως ε, ε, στις χώρες που έχει παρέμβει δεν χαίρει μεγάλης εκτιμήσεως. Η συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ε, μπορούσε να είναι χρήσιμη. Σημείωσα την ημερομηνία που αναφέρατε για την ε, ε, συνάντηση σας του χρόνου με τον κύριο Ρούντι Τάλερ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα είμαστε σε επαφή. Μόλις λοιπόν θα μας το επιτρέψει το πρόγραμμά μας με τα μεγάλης χαράς θα σας επισκεφθούμε στην οργάνωσή σας στη Γενέβη και παραμένουμε στη διάθεσή σας. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, το τηλέφωνο μας είναι γνωστό. Εν ονόματι του ΕΛΚ και προσωπικά σας διαβεβαιώ ότι προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία με την οργάνωσή σας. Ο κύριος Θέρκας και μετά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και, μένα, και, και εγώ θα καλωσορίσω τον κύριο Ράιντερ Και πρέπει να πω ότι εκφράζω και αισθήματα ηρεμία και φυσικασμού, διότι έφυγε ο κύριος Σοναρίβα, ο οποίος ήταν ένας φίλος, αλλά ήρθε άλλος. Και δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι η Γενική Γραμματεία της ΔΟΕ βρίσκεται σε, στα καλύτερα χέρια. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική και παραγωγική μεταξύ ημών. Για τις ε, αξίες και τους στόχους θα ήθελα να συγκρίνω την τροχιά των δυο μας οργανώσεων. Όλα αυτά μου φαίνονται μια αγγελική μουσική. Βρίσκομαι στον παράδεισο Βλέπουμε ότι σήμερα στην κοινωνία οι αξίες έχουν παραμεριστεί, τα πάντα έχουν ε, αντικατασταθεί από το κέρδος, από την παραγωγικότητα. Ε, έχουμε την αίσθηση ότι μας οδηγάνε με ένα αυτοκίνητο και δεν κοιτάνε ποτέ πίσω το δρόμο, την ιστορία που έχουμε πίσω. Και επειδή δεν κοιτάνε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάνε μόνο μπροστά και χωρίς να κοιτάνε πίσω, μας ταράζουν στις γωνίες και για στη σύμπτωση κοιτάνε μόνο δεξιά. Και αυτό συμβαίνει διότι βρισκόμαστε στα χέρια αυτών των αρχηγών, όπως είπε κάποιος, έχουμε τη, τη μεγαλύτερη κρίση μετά τον, το, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βρισκόμαστε στα χέρια της χειρότερης αρχηγίας, της χειρότερης leadership μετά <coughs> τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς λοιπόν ταινίζουμε προς τη Γενέβη όπως γινόταν το 1920 οι εργάτες, οι Έλληνες εργάτες, οι Ισπανοί εργάτες συνεχίζουν να έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. η οποία Ευρώπη βέβαια δεν είναι μεταξύ των καλύτερων μαθητών, διότι αρχίζει και αυτή και ξεχνάει τα διδάγματα της ιστορίας. Έχω μία ερώτηση συγκυριακή. Πρώτον, απασχόληση. Διάβαζα εχθές την έκθεση για την κατάσταση της απασχόλησης στον κόσμο το 2012. Μπράβο, μπράβο. Διότι κοιτάτε την πραγματικότητα κατάφατσα και αντιπροσωπεύεται δηλαδή ε, πάρα πολύ καλά την, ε, την κατάσταση. Λέτε χωρίς η λιτότητα δεν φτάνει, χωρίς ανάπτυξη δεν γίνεται τίποτα. Ρωτώ λοιπόν, αυτή η παγίδα της λιτότητας που μειώνει την ποιότητα της απασχόλησης, ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Είδατε εσείς τι γίνεται με τις εκθέσεις της Τρόικας που πάνε στο νότο της Ευρώπης. Αυτά τα κείμενα της Τρόικα δεν αντιβαίνουν με αρχές της ΔΟΕ. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι ούτω ώστε η ΔΟΕ όχι μόνο να προστατεύει τους Ινδούς ή Κινέζους εργάτες που βρίσκονται μακριά, αλλά και τους Ευρωπαίους εργάτες δίπλα στο σπίτι μας. Τώρα, κοινωνική συνοχή, πολύ σημαντικό θέμα, λόγω ιστορίας και τροχιάς. Εμείς ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα λόγια δεν σημαίνουν τίποτα ή σημαίνουν το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλουν να πούν. Λοιπόν, εδώ ακούγεται συνέχεια να μεταρρυθμίσουμε το κοινωνικό μας σύστημα. Μα εδώ δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, πρόκειται για αντιμεταρρύθμιση. Τι πιστεύετε εσείς για αυτές τις πλατφόρμες, για τα ελάχιστα κοινωνικά δεδομένα. Λοιπόν, τι θα γίνει με το social protection floor, με τον συμβιβασμό της ΔΟΕ. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να λύσουμε με την ευρωπαϊκή ατζέντα σωστές, Κατα... σωστές θέσεις για να ξεπεράσουμε καταστάσεις δύσκολες, ε, για να μην μείνουμε εμείς ε, απροστάτευτοι σε αυτήν την κατάσταση αδικίας και ψευδορισμού που μας καταλαμβάνει. Θα αφήσω όλους ε, να εξαντλήσουν το, να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους γιατί αυτό είναι σημαντικό σε μια τέτοια ε, θεματική αλλά θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο να μπορέσει να μιλήσει και ο εισηγητής. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Ράιντερ εκπροσωπώ τους φιλελεύθερους εδώ και είμαι ε, Ιρλανδή. Καταρχήν σας καλωσορίζω εδώ διότι είχα συνεργαστεί ε, και γνώριζα τον προκάτοχο της θέσεώς σας και χαίρομαι που σας γνωρίζω και ε, σας. Όπως είπατε η Διεθνής ε, Οργάνωση Εργασίας έχει υπάρξει πολύ χρήσιμη και μας έχει βοηθήσει εξού και αναγνωρίζεται το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλές φορές όμως έχουμε τόσες που δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Είπατε ότι χρειαζόμαστε μία δημοσιονομική ε, βελτίωση και είπατε ότι σε ορισμένες ε, κυβερνήσεις δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις και αυτές που έχουν τους πόρους δεν επενδύουν επαρκώς. Επίσης πρέπει να βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, βλέπω ότι γίνεται π.χ. στην Ιταλία που είναι τραγικό. Δηλαδή αν σκεφτείτε τι γίνεται δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε και ε, τι θα γίνει, πώς πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους μας. Διότι στην ε, Ιρλανδία μόλις έχουμε ε, ε, προσυπογράψει ένα δημοσιονομικό σύμφωνο. Ήθελα να ρωτήσω, εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, υπάρχει κάποια πρόοδο στην οποία πιστεύετε ότι μπορείτε να επιτύχετε, διότι μιλήσαμε προηγουμένως για το ψήφισμα και για το γεγονός ότι μπορεί κανείς να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις ε, της κρίσεως. Θα ήταν λοιπόν καλό να ξέρουμε ότι έχουμε κάποιον ο οποίος μας ακούει. Και υποθέτω ότι το τελικό μου ερώτημα είναι ότι αν δείτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία αλλά και στη Γερμανία και στην Πολωνία και στη Φιλανδία και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ρήξη, ένα σχίσμα στην Ευρώπη μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί αλλού και αυτό πρέπει όμως να περιλάβει και την ε, Ελλάδα και την Ιρλανδία και ε, δεν έχει ακόμη γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για ένα κοινό πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε και εντάθηκε από το θέμα του κοινού νομίσματος. Ό,τι και να είναι, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, οπότε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την αλληλεγγύη η οποία χρειάζεται, η οποία δεν σημαίνει εγώ έχω δίκιο και εσύ άδικο, αλλά να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Σας έχω κάνει ερωτήματα που ίσως σας φαίνονται αδύνατα και σας παρακαλώ αν μπορέσετε να μου απαντήσετε σε ό,τι μπορέσετε. ο Τόμας Χάντελ και μετά ο Τόμας Μαν. Καταρχήν, ε, κύριε Γενική Διευθυντά, ε, σας συγχαίρω για την εκλογή σας. Ε, βλέπω ότι και οι δύο είμαστε από το συνδικαλιστικό τομέα, το διάβασα στη βιογραφία σας και αυτό είναι πολύ καλό και έχω τρεις σύντομες και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πέρυσι όταν επισκεφτήκαμε στη, τη Γενέβη μπορέσαμε να δούμε πώς κινείται η Διεθνής Οργάνωση Εργασία για να υπάρχει ένα κοινωνικό βήμα, ένα πρότυπο κοινωνικής ασφάλισης για διάφορα κράτη και το βήμα το κοινωνικό είναι χαμηλότερο σε αναδιόμενες χώρες από ό,τι αλλού. Οπότε ε, πόσο έχει προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, πότε μπορείτε να το παρουσιάσετε και ε, να εμπλέξετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης στη συνέχεια της κρίσεως αυτές ε, και των πολιτικών λιτότητων όχι μόνο σε χώρες εκτός ε, Ευρώπης βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη καταλύονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα το είδαμε στην Ουγγαρία το είδαμε με την αντιμετώπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Ιταλία οπότε υπάρχει μια τοποθέτηση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας εν τω μεταξύ ε, ε, ε, είστε εδώ στην Ευρωπαϊκή στην Επιτροπή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά η φωνή σας δεν ακούγεται πέραν αυτής της Επιτροπής. Η οργάνωσή σας ε, τι κάνει για να προβάλλει περισσότερο το έργο της στο Κοινοβούλιο κατά τρόπον ώστε όταν καταρτίζονται ε, οδηγίες να μπορεί κανείς να εφαρμόζει και περισσότερες αρχές της διεθνούς οργανώσεως εργασίας εργασίας. Ο κύριος Τόμας Μαν. Και εγώ θέλω να, σα να σας συγχαρώ, ίσως αντιληφθήκατε ότι είμαι Γερμανός. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι ο φυσικός συνέτερος όχι μόνο της Επιτροπής μας αλλά και του Κοινοβουλίου και πάντοτε στα ψηφίσματα ε, που θεσπίσαμε υπήρχε ευρεία αποδοχή και δεν ήταν ψεύτικη. Ε, δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Πρέπει λοιπόν να καλύψετε το κενό, το μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει μεταξύ ε, της ε, σημερινής κατάστασης και του μέλλοντος και ιδίως ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η μελλοντική εξέλιξη. Και αν μιλάμε για κρατικό σύμφωνο ή δημοσιονομικό σύμφωνο, βεβαίως δεν θέλουμε να καταργούνται και να καταλύονται τα εργατικά δικαιώματα αλλά ε, η δημοσιονομική, το δημοσιονομικό σύμφωνο δεν είναι ένα στόχος, είναι μία ανάγκη η οποία είναι επιτακτική κατά τρόπον ώστε να υπάρξουν ε, τα αναγκαία μέτρα για εξοικονόμηση πόρων που θα μπορέσουν να επενδυθούν. Εσείς ε, τι μπορείτε να προσφέρετε διότι πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη στις κινήσεις του και την προοπτική τη μελλοντική. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μπορεί να διαφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο θέσεων και να μας εξηγήσει ότι αυτές οι πορείες πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση για να αποφύγουμε να περιθωριοποιούνται οι άνθρωποι και εργαζόμενοι. Επίσης ακούσαμε για τις προσπάθειές σας στην Ασία και στην Αφρική να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας. Τι γίνεται όμως με την Κίνα, ε, διότι θέλουμε να υπάρχει κοινωνικό σύμφωνο και έχουμε παράπονα πολλά για την Κίνα όπου μας λέγουν ότι δεν υπάρχουν πλέον κοινωνικά δικαιώματα ή ε, ε, εκπρόσωποι ε, των χωρών που αντιμετωπίζουν κρίση και είναι σε στασιμότητα δεν μπορούν, λέγουν ότι δεν μπορεί κανείς να κινηθεί αν δεν ρωτήσει την άδεια των δημοσιονομικών αρχών. Υπάρχει δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές κάποια εμπλοκή της Διεθνούς ε, Οργανώσεως Εργασίας επεμβαίνεται και στην Αφρική, στις δικτατορίες ή στην Κίνα. Ε, ξέρω ότι πρέπει να προστατεύσει κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα. Σωστά είπατε ότι είναι παίκτη κλειδί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω όμως οι παίκτες μας να αρκούν. Πολύ ωραία. Η Γιούτα Σάιλοκ. Ευχαριστώ. Το κύριε Πρόεδρε ε, και εγώ θέλω σαν συνδικαλίστερα να ε, συγχαρώ τον συνδικαλιστή. Ε, ερωτήσεις. Καταρχήν όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή αγορά πώς είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος διότι βλέπουμε ότι άλλες περιοχές διεθνώς ε, είναι φτηνότερες και γι' αυτό υπάρχει μία μετατόπιση ε, βιομηχανικών θέσεων εργασίας για να μπορέσουν να επιβιώσουν τι θα γίνει στην Ευρώπη μπορούμε να δεχτούμε οι θέσεις αυτές στο μέλλον να εξαφανιστούν ή θα πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς σε, αυτή, ε, την, ε, σε αυτό το διαγωνισμό υποτιμήσεων. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο μας λέγεται ότι η και οι συνθήκες εργασίας πρέπει να γίνουν πιο ελαστικοί και πιο ανταγωνιστικοί. Ερώτησης. Ε, ε, ε, δεν δεν θα έπρεπε κανείς να δει τι γίνεται στην Ευρώπη πρώτα και μετά να τη συγκρίνει στο εξωτερικό. Ποιοι είναι δηλαδή οι, ε, τα σημεία συγκρίσεως και οι χώρες συγκρίσεως που θεωρείται ότι είναι πιο ανταγωνιστικές από την Ευρώπη. Ε, επίσης έχει λεχθεί πολλές φορές ότι η έλλειψη κατωτάτων μισθών και κατά των ορίων μισθών οδηγούν πολύ συχνά σε προσωρινές θέσεις εργασίας και ε, στα, στις περιπτώσεις αυτές έχουν ε, επιπτώσεις και στις μελλοντικές ε, εξελίξεις διότι τι θα γίνει και πώς αυτή η κατάσταση θα έχει επιπτώσεις σε άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Ευρώπη. Οι διερμηνείς μέχρι τις 12.30 θα είναι εδώ. Τόσε ερωτήσει σε 7,5 λεπτά, πού να τέλος θα προσπαθήσω να είμαι σωστός σε όλους αυτούς που κάνουν τον κόμμα να τέλο. θα προσπαθησω να ειμαι σωστό σε όλου αυτού που κανουν τον πρώτα σας ευχαριστώ και πάλι ε, για, για αυτή τη θετική σα ε, υποδοχή, για τον ενδιαφέρον σα. και όταν θα βγαίνω αυτή την αίθουσα θα είμαι πιο, πιο αισιόδοξο, όχι γιατί έχω βρει με θαυματουργό τρόπο τις λύσεις για όλα τα προβλήματα τα τελευταία 45 λεπτά, αλλά γιατί προβληματιζόμαστε να αναζητούμε μια λύση που μπορούμε να τη βρούμε από κοινού. Μια γενική παρατήρηση που θέλω να σας πω σε σχέση με τη συζήτηση αφορά αυτό το, τη, γενικότερη κατάσταση ε, που το είχατε και εσείς σε ερωτήσεις σας ε, όλες υπόψη και διαφορετικούς τρόπους μιλήσατε πολύ, πολύ από σας σχετικά με αυτό ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία, τα οποία φαίνονται τόσο εντυπωσιακά. Το όπως είπε και ο συνάδελφος από την Ισλανδία. Πού να ξεκινήσει κανείς. Ε, το συγχωρείτε μπορεί να γίνει κανένα να σταυρώσει τα χέρια να, να τον πιάσει παράλυση, να μην κάνει τίποτα. Και το θέμα είναι, δεν το λέω για πραγματικότητα, λέω για την αντίληψη, την αντίληψη του πώς αντιμετωπίζεται η κρίση προσοχή, η γενική εντύπωση επομένως είναι ότι υπάρχει άδικη αντιμετώπιση, ότι το βάρος έχει κατανεμηθεί άνισα και ότι η ρίζα του κακού ξεκινάει από κέντρα εξουσίας από τον οποίο δεν έχει κανένας. Δεν έχει ο κόσμος τουλάχιστον έλεγχο. Επομένως, εσείς τώρα καλείστε να βγάλετε το φύριο από την τρύπα και όπως είπατε σωστά, είμαστε όπως είμαστε τώρα, όμως σε μας απόκειται να, ε, να, να, να, να, βρούμε την, την διέξοδο στο τούνελ, την έξοδο και μου αρέσει που είμαι εδώ γιατί κάποτε και εγώ ήμουν σε ένα χώρο τέτοιο, όντως πρόκειται περί και βλέπω όμως ότι υπάρχει θέληση να βρούμε την, την, την διέξοδο. Και αυτό είναι τρομερή ενθάρρυνση τώρα σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που ρωτήσατε. Όντως το θέμα της απασχόλησης είναι υψίστη προτεραιότητα. Και στην διάσκεψή μας μιλήσαμε ε, στη ΔΟΕ για την ε, ανεργία των νέων και είπαμε ότι το να μπορούν να βρουν οι νέοι μια αξιοπρεπή δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ για κάποιους που βρίσκονται στα μέσα της τρεις δεκαετίας της ζωής τους και δεν έχουν ποτέ βρει θέση, δεν έχουν ποτέ βρει δεν έχουν βρει θέση στην αγορά της απασχόλησης. Οπότε θα πρέπει τελικά να δούμε ότι για το, για το κάθε τέτοιο πρόσωπο πρόκειται για ένα δράμα, μια τραγωδία. Είναι κοινή μας ευθύνη αυτή και να βρούμε μια απόκριση. Οπότε να, αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει για να αναζητήσουμε τη λύση. Τώρα όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική προστασία. Πολλές ερωτήσεις, η ιδέα διάσκεψη της ΔΟΕ ε, ψήφισε μια, ένα, ένα, ένα, μια σύσταση ε, και επομένως τώρα έχουμε ένα όργανο, δεν είναι δεσμευτικό, ε, το οποίο ε, επιδέχεται κύρωση, το οποίο αποτελεί βέβαια συμβουλευτικό απλώς εργαλείο για το τι μπορεί να γίνει από πλευράς κοινωνικής πρόνοιας παντού και επίσης αποτελεί για ένα λιθαράκι για την προσπάθεια του, του G20. Δηλαδή, όπως είναι σήμερα η κατάσταση, μόνο 20% 100 από τους εργαζομένους έχουν πρόσβαση σε, σε, κάποιο είδους κοινωνική πρόνοια. Και τα, στατιστικά λένε ότι χρειάζεται επίστευτη επένδυση ούτως ώστε να, έχουν, ε, να έχει ο κόσμος όλος ε, κάποιο είδους κοινωνική πρόνοια. Όχι, όχι, δεν είναι το ίδιο στην Μπαγκλαντές όπως και στο Μπραζίλ, στη Βραζιλία, αλλά το να κάνουμε αυτή την κίνηση θα αλλάξει τη ζωή πραγματικά τόσων εργαζομένων. Όλα αυτά επομένω είναι προτεραιότητά μας και θα τα παρακολουθήσουμε. Επίσης, δικαιώματα συνδικαλιστών, δικαιώματα εργαζομένων, όλα αυτά καταπατούνται παντού και το Global Jobs Pact του 2009 θεώρησε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και είπαμε ότι αυτό δεν είναι θέμα κάποιου κόμματο, αλλά είναι κάτι που αφορά όλα τα συνδικάτα, όλε τι κυβερνήσει. Και είναι απαράδεκτο αυτό, δεν είναι, δεν είναι απόκριση στην κρίση. Ε, ούτε, ούτε ο ξεφτελισμός των μισθών αποτελεί λύση. Να οι θέσει τη ΔΟΕ. Όντως, καταποντούνται τα δικαιώματα και να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί πολλές φορές έχουμε πει και εμείς ότι σε μερικές φορές, σε μερικές περιστάσεις, όντως έχουμε καταπάτηση δικαιώματα με την κρίση, αλλά, αλλά και πολλούς αποσχολεί αυτό. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι δίνουν ως αντάλλαγμα την παρέτηση από τα δικαιώματά του για να μείνουν στη δουλειά. Αυτό δεν είναι καταπάτηση δικαιωμάτων. Ας είμαστε προσεκτικοί για το τι διατυπώσει κάνουν. Τώρα όσον αφορά την ε, πολιτική απασχόληση στη Γερμανία δεν μπορώ τώρα να μπω σε, αυτό το, το, σε αυτή τη συζήτηση αλλά το ατού της Γερμανίας είναι τα θεσμικά όργανα και η κουλτούρα του διαλόγου. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν πια στη Νότια Ευρώπη. Είναι μια από τι τραγωδίε τη Ελλάδο ότι ο κοινωνικό διάλογο έχει φρενάρει και ότι τα θεσμικά όργανα εκεί χωρίς να ήταν ποτέ σπουδαία τώρα είναι σε τραγική κατάσταση και γι' αυτό και στην Ελλάδα θα δούμε δράματα όχι μόνο από πλευράς μισθολογικού αλλά και από πλευράς θεσμικής. Για την Κίνα τώρα. Όχι, όχι, δεν είναι καλοπιστικά. Δεν είναι προς το Θεαθήνε μόνο αυτές οι κινήσεις της Κίνας. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι Όντω, από το βράδυ στο πρωί δεν είναι δημοκρατία εκείνα, Όμω, η καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι του, του σούπερ εξαγωγέα. Αυτό το πιστεύω να κάνουν είναι ξαφνικά, που δεν το κάνανε παλιά, να κάνουν τον κόσμο να αποταμιεύει για να μπορεί να έχει και εσωτερική αγορά ισχυρή. Ε, ή έχουν μακρά διαδρομή μπροστά του. Και ε, ήθελα να πω ότι υπάρχει κάποια πρόοδο. Δεν είπα εγώ ότι υπάρχει μια τρομερή πρόοδο. Πολλά, πολλά μπορούσα να πούμε. Όμω, όμω, εν κατακλείδη, θέλω να σα πω δύο λόγια, δύο λόγια τα οποία ε, είπε ο ισπανό συνάδελφο είπε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε κοινικοί στο τι θα κάνουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο κανεί να πέσει στο, στον κινησμό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Άρα, έχουμε μεγάλη ευθύνη, υπευθυνότητα. Δεν είναι δυνατόν να γινόμαστε κοινικοί. Η λέξη κλειδί τώρα είναι αλληλεγγύη. Μα αφορά όλου. Τα προβλήματα δεν είναι ούτε ατομικά ούτε ιδιωτικά. Είναι κοινά. Και αυτό αφορά επομένω όλο το πολιτικό φάσμα, αυτό που λέω. Αυτό είναι μόνο η αρχή των όσων έχουμε να πούμε. Σας ευχαριστώ με καλέσατε. Δώσε ευκαιρία να σας ακούσω και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας τους αμέσως επόμενους μήνες. Εγώ ωφελούμαι από αυτό και, και η ΔΟΕ και ελπίζω και εσείς. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι, θίξατε διάφορα τα οποία συζητήσαμε. Δεν είπαμε για την ανεργία, αλλά ξέρετε, η ανεργία μας απασχολεί πάρα πολύ βέβαια και τι να σας πω. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι σε τέσσερις μήνες ο νέος που κάνει τη δουλειά του ή θα μπαίνει σε κάποιο στάζ ή θα βρίσκει κάποια δουλειά ή τέλος πάντων θα ξαναμπαίνει στην κατάρτιση στην εκπαίδευση Και σήμερα το πρωί μόλις ψηφίσαμε έκθεση που ακριβώς ζητούμε από την Κομισιόν να κάνει αντίστοιχα. Επίσης αναφέρατε τα θέματα της αξιοπρεπούς εργασίας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει και αξιοπρεπής αμοιβή, μισθός, μέσα στη Γερμανία. και ε, το, η αγορά εργασία τη Γερμανία είναι βασικό θέμα, πρέπει και εκεί να στρέψουν την προσοχή μας. Επίση για την Κίνα, πάλι. Και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προσέξουν την εσωτερική τους αγορά. Να σταματήσουν να είναι έτσι ένα εργαστήρι που παράγει για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Άλλαξαν τα πράγματα μας και, και, γι' αυτό και νομίζω ότι και ΔΟΕ. Και βεβαίω αυτό είναι καθήκον σας να βρείτε μια λύση. Και είναι και εδώ πέρα διακύβευμα και οι συντάξεις. Και γι' αυτό ακριβώς και θα πρέπει να έχουμε περισσότερη συνέπεια στην πολιτική μας. Γιατί ξαναρχίζουμε τώρα στην αφετρία της ζήτησης. Καλά, καλά, θα, θα, θα, τα πούμε και άλλη φορά, θα, συνεχίσουμε. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα θα είναι στις... Ε, θα ξαναπούμε στις 12 Νοεμβρίου. Και οπωσδήποτε, επί τη βάση των όσων ενδιαφερόντων μας είπατε τώρα, θα... Ε, και τότε θα σας πούμε πώς και πώς Τέλο πάντων, ελπίζουμε ότι θα έρθουν εδώ πέρα τα, τα στελέχη της Επιτροπής μας να σας ακούσουν.